Okay, so let me open, uh... Ωραία, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίσω την έναρξη της συνεδριάσεως. Είμαστε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Και με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω εδώ 16 βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια από 9 χώρες μέλη με άλλους αξιωματούχους, 40 συνολικά από τα Εθνικά Κοινοβούλια, για να ανταλλάξουμε απόψεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2019. Είναι μια πολύ σημαντική για να έχουμε συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, γιατί έχουμε και τις ε, συστάσεις αναχώρα που εγκρίθηκαν πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές από το Συμβούλιο. Και τώρα πιστεύουμε ότι θα τεθούν σε εφαρμογή με νομοθεσία. Επιπλέον, έγινε συζήτηση σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια και πιστεύουμε ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο και σε άλλες χώρες. Είναι καλό λοιπόν να συζητήσουμε μαζί τον κύκλο αυτό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2019. Τώρα υπάρχει και έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας η οποία ολοκληρώνεται τώρα στην δικιά μας Επιτροπή με εισηγήτρια την κυρία Ντελάνγκη από το ΕΛΚ. Στόχος μας σήμερα είναι να συζητήσουμε τις τροπολογίες. Υπάρχουν 272 τροπολογίες και θα ψηφίσουμε για αυτές τις 2 Οκτωβρίου στην Επιτροπή μας. Τώρα, μερικά πρακτικά ζητήματα. Έχουμε 23 γλώσσες στη διάθεσή σας, οπότε μπορείτε να διαλέξετε. Επίσης, υπάρχουν κάρτες για ομιλία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφόσον θέλετε να ζητήσετε να παρέμβετε. Θέλετε να πάρετε μέρος στη συζήτηση. Αν ένας ε, ε ευρωβουλευτής θέλει να μιλήσει, επίσης να συμπληρώσει την καρτέλα. Τώρα, γενικά, χρόνος ομιλίας. Έχουμε δύο ώρες συνολικά και έχουμε αποφασίσει ότι θα ξεκινήσουμε με τους σκιώδες εισηγητές, μετά θα έχουμε δύο εκπροσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και μετά έναν Ευρωβουλευτή. Η κάθε παρέμβαση πρέπει να περιοριστεί το πολύ στα τρία λεπτά. Και αν χρειαστεί θα προσαρμόσουμε τους κανόνες ε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Εστερντελάνγκια, αλλά η Εστερντελάνγκια δεν είναι εδώ ακόμα. Έχει αντικατασταθεί από τον κύριο Μπέργκερ από το ΕΛΚΑ που θα παρουσιάσει τελικά τις παρατηρήσεις της κυρίας Ντελάνγκια και μετά θα έχουμε τα Εθνικά Κοινοβούλια. Λοιπόν, έχετε το λόγο κύριε Μπέργκερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε δύο εκθέσεις. Έχουμε, πήραμε την πρώτη έκθεση ε, τώρα όμως είναι η φορά, είναι η στιγμή για να καταθέσουμε την δεύτερη έκθεση που αναλύει τις ε, ειδικέ ανασυστάσεις χώρα. Αυτές οι CRAs, όπως λέγονται, εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο πριν από το Κοινοβούλιο. Αυτές οι ειδικέ ανασυστάσεις χώρα ε, συμβουλεύουν τα κράτη-μέλη το πώς να αυξήσουν τις θέσεις απασχόλησης, τις επενδύσεις ε, και παράλληλα να διατηρήσουν υγιή δημόσια οικονομικά. Ας δούμε λιγάκι ποια είναι η οικονομική κατάσταση. Η θετική οικονομική τάση προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί ε, βέβαια σε χαμηλότερο ρυθμό. Στις κοινωνίες μας παραμένουν σημαντικές προκλήσεις και για τις οικονομίες κοινωνίες μας εξακολουθεί να είναι υψηλή η ανεργία των νέων. Η οικονομική κίνδυνη και η ε, πολιτική ανασφάλεια δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις. Αντιμετωπίζουμε όλο και μεγαλύτερη παγκόσμια ανασφάλεια λόγω του εμπορικού πολέμου με την Κίνα και υπάρχουν και εσωτερικοί κίνδυνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του Brexit. Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει χαμηλές προοπτικές ανάπτυξης σε σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να ε, βασιστούν στην πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία έτη, ακολουθώντας ε, μια σωστή δημοσιονομική πολιτική, εφαρμόζοντας ε, μεταρρυθμίσεις ε, και ακολουθώντας ε, σωστές ε, στρατηγικές, αυτά ως πηξίδα για τον εξυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ε, Υπεύθυνε σε δημοσιονομικές πολιτικές και συμβατότητα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αυτά χρειάζονται για να έχουμε ανθεκτικές οικονομίες που θα είναι θωρακισμένες για την επόμενη ύφεση και θα είναι και θωρακισμένες απέναντι στις κοινωνίες, τις γυράσκουσες κοινωνίες. Ε, τα, ε, τα δημόσια χρέη, ε, το δημόσιο χρέος κρατών που είναι πάνω από το ΑΕΠ, αυτό μπορεί να οδηγήσει ε, στο να περιστεί ανάπτυξη τα επόμενα έτη. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχουν διαρθρωτικέ ε, μεταρρυθμίσει για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να έχουμε περισσότερες αντεκτικές οικονομίες. Η αγορά εργασία του 21ου αιώνα απαιτεί επενδύσεις ε, σε δεξιότητε σε παιδεία και ε, διαβίου μάθηση. Οι οικονομίε ε, θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν την ύφεση. Αυτό απαιτεί ευέλικτη αγορά εργασία, ε, ανταγωνιστικέ αγορέ προϊόντων, ποιοτικού θεσμού και αποτελεσματικό σύστημα δικαιοσύνη. Όλα αυτά αποτελούν απαιτούν και ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν επενδύσεις για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα, οι δεξιότητες, η καινοτομία και παράλληλα να βελτιωθεί και το δυναμικό ανάπτυξης. Υπογραμμίζουμε ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν και άλλα μέτρα για να αντιμετωπιστεί το χάσμα επενδύσεων στην Ευρωζώνη που έχει σωρευτεί από τότε που ξέσπασε η ε, κρίση. Βέβαια υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η υποστήριξη των δημόσιων και των ιδιωτικών ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό ε, πρέπει να ε, λάβει χώρα έχοντας πάντα κατά νου ε, το ΑΕΠ. Η δική μας δουλειά λοιπόν τώρα είναι να αναλύσουμε το περίφημο φαύλο τρίγωνο για να μπορούμε να πούμε στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τι κατά τα άποψή μας είναι σημαντικό και ποια είναι η απαραίτητη πολιτική καθοδήγηση για το μέλλον. Νομίζω σε γενικές γραμμές ε, αυτά είναι τα βασικά θέματα. Άκουσα ότι η επόμενη ε, συνεδρίαση των ε, σκιωδών θα γίνει αύριο και εκεί ε, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε περαιτέρω τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστούμε και για την ε, αντικατάσταση. Να δώσω το λόγο στον πρώτο εθνικό βουλευτή από το Ρουμανική Γερουσία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο έως τρία λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πω δύο λόγια στα Ουγγρικά, γιατί εδώ εκπροσωπώ και τους Ούγγρους στην Ρουμανία, αλλά και ε, την γερουσία της Ρουμανίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο Γιώζεφ ε, Άντελ είναι ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα και θα περάσω τώρα στα αγγλικά. Είναι πολύ σημαντικό το ευρωπαϊκό οικοδομήμα. Όπως ξέρετε η Ρουμανία συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Εκτιμούμε τη σημασία που δίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Κομισιόν ε, στον ενδυνάμωση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών ε, και το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη και του σχετικού στόχου. Ε, σε ό,τι αφορά την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη για το 2019, θεωρούμε ότι υπάρχει συνεκτική προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διατηρηθούν οι τρει κυρίε προτεραιότητε. εξηγεσμένα οικονομικά, επενδύσει σε υψηλού επίπεδου και μεταρρυθμίσει που θα επικεντρώνονται σε αυξανόμενη παραγωγικότητα, συμμετοχή και θεσμική ποιότητα. Δεδομένων των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, η αξιολόγηση των επενδυτικών αναγκών υποστηρίζει τις προσπαθίες μας στο να θέσουμε τις σχετικές προτεραιότητες για την επόμενη δεκαετία. Αυτή η αξιολόγηση επίση αποκαλύπτει τον τρόπο που τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής μπορούν να συνεισφέρουν σχετικά. Επομένως, η ανάλυση που περιλαμβάνεται στις εκθέσεις αναχώρα συνεισφέρει σημαντικά για να έχουμε ένα καλύτερο συσχετισμό του προγραμματισμού των κονδυλίων με τα διάφορα στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και αποτελεί τη βάση του διαλόγου των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της Συμφωνίας Εταιρική Σχέσης. Αναμφισβήτητα, καλύτερα στοχευμένε επενδύσει θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου η άποψή μα είναι ότι μέσω πρόθεσμα θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην εφαρμογή περισσότερο παρά στο να έχουμε περαιτέρω διαδικασίες εργασία. Η Ρουμανία θα ανταποκριθεί με μέτρα που θα επιβεβαιώσουν την πολιτική βούληση να συνεχίσουμε τι μεταρρυθμίσει που συνεισφέρουν σε βιώσιμη και συμμετοχική ανάπτυξη στο να έχουμε αυξημένη αποτελεσματικότητα επενδύσεων και απασχόληση υψηλή ποιότητα. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σας ευχαριστώ κύριε Αντάλ για την παρέμβασή σας και για τη δέσμευσή σας και την αφοσίωσή σας. Ο κύριος Κόκος επίσης από τη Ρουμανία, από το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ρουμανία συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και εκτιμάται πόση σημασία δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το εργαλείο το οποίο θέλει να ενδυναμώσει τι κοινωνικέ, οικονομικέ, πολιτικέ τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και του στόχου του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά την ετήσια ε, ανάπτυξη, εμεί εκτιμούμε την προσέγγιση τη Κομισιόν που αναφέρεται στι τρει κύριε προτεραιότητε, τα δημόσια οικονομικά, τα εξηγιασμένα στις, επενδυ... στις υψηλές ε, ποιότητες επενδύσεως και στην αύξηση της ε, παραγωγικότητας, στην συμπερίληψη και τη θεσμική ποιότητα. Επίσης, χαιρετίζουμε την πρόσφατη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που αφορά ε, την πρόθεση των επενδύσεων ε, και τις διαρθρωτικές επενδύσεις που και σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη έχοντας κατά νου τις διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την αξιολόγηση των επενδυτικών αναγκών. Αυτή υποστηρίζει τη δική δική μας ανάλυση για την επόμενη δεκαετία και τις σχετικές προτεραιότητες ε, και το πώς μπορούν τα κονδύλια συνοχής να συνεισφέρουν. Επομένως, η ανάλυση των ε, ε, εκθέσεων αναχώρα συνεισφέρει στο να προγραμματίσουμε καλύτερα τα διάφορα στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και αποτελεί τη βάση του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη προετοιμασία τη Συμφωνία Ιστορική σχέση. Έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο για το να εντοπίσουμε ε, τι εθνικέ προτεραιότητε για να αναπτύξουμε επενδυτικέ πολιτικέ. Ε, πιο στοχευμένε επενδύσει θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη του στόχου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θεωρούμε κατάλληλη την προσέγγιση τη Κομισιόν, ε, η οποία προβαίνει σε ειδικέ ανά αναχώρα και θέτει προτεραιότητε θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην εφαρμογή και όχι στην εισαγωγή κάποιων ε, πρόσθετων ε, έργων. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις που να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, στη βιωσιμότητα και στην συμπερίληψη. Πρέπει να έχουμε υψηλή ποιότητα σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Ο πρώτος Ευρωβουλευτής που θα πάρει το λόγο είναι η σκιώδηση εισηγήτρια από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Παρακαλώ, η κυρία Λαλίκ. Ευχαριστώ πολύ. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο κάνει συστάσεις αναχώρα προκειμένου να ενισχυθεί ανάπτυξη για απασχόληση και να καταπολεμηθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Όταν σήμερα κοιτάμε τα μακροοικονομικά στοιχεία, διαπιστώνουμε ότι από το 2011 μέχρι σήμερα, όσον αφορά την ανάπτυξη, που ήταν υποτονική, αδύναμη, δεν ξεπερνάει το 1,2 ή 1,5% το πολύ τα καλύτερα χρόνια, ότι υπάρχουν μακροοικονομικές ανισορροπίες, κυρίως όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο, τόσο μέσα στην Ευρωζώνη όσο και εκτός, και ε, μία ανεργία που είναι 7,5% περίπου κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε με τα 87 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι ζουν στα όρια της στόχιας. Επίσης διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετές επενδύσεις στην Ευρωζώνη. Είναι κάτι το οποίο λέμε και ξαναλέμε όλοι οι οικονομολόγοι, το Δούνου του, ο, ο ΣΑ κλπ και ότι 24 από τις 28 χώρες τα 10 τελευταία χρόνια δεν έκαναν αρκετές επενδύσεις, ούτε καν αρκετές για να μπορέσει κανείς να προστατεύσει την ε, κληρονομιά του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο απολογισμός δηλαδή δυστυχώ δεν είναι θετικό, ενώ υπάρχουν και άλλε προκλήσει μπροστά μα, όπω είναι η κλιματική απορρίθμιση με την άνοδο τη θερμοκρασία, Εξού και οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτε που εκπροσωπώ εδώ σήμερα θέλουν το κείμενο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να περάσει από διαπραγμάτευση στην Επιτροπή μας για να του δώσουμε νέα πνοή. Να λάβουμε υπόψη μας τους περιβαλλοντικούς και τους κοινωνικούς δείκτες. Το θέμα επίσης της ενεργειακής φτώχειας που αφορά 5 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη μας και να ξαναδούμε την οικονομική και κοινωνική πολιτική ε, μέσα από το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, να δούμε τι γίνεται με τις επενδύσεις που έχουν σταματήσει. Πώς θα πετύχουμε την οικολογική μετάβαση ώστε να δημιουργηθούν εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, κάτι το οποίο ζητάει το Ευρωπαϊκό Εξήμενο. Θέλουμε λοιπόν μεγαλύτερη ευελιξία στον τομέα ε, του συμφώνου, το οποίο είναι υπερβολικά αυστηρό απέναντι στις οικονομίες μας. Ε, γίνονται ε, αλλαγές σε διάφορου τομεί, όχι μόνο στο περιβάλλον, στην ψηφιοποίηση και όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στην έκθεση, όπω επίση η πολιτική κατάρτιση και εκπαίδευση, οι εγγύσει για τα συστήματα κοινωνική ασφάλισης, η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στι διαπραγματεύσει. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για μα. Θέλουμε επίση αναρμόνιση τη Ευρωπαϊκή φορολογία, ώστε οι χώρε μέλη να έχουν περισσότερα μέσα στη διάθεσή του και να πάψει αυτή η κούρσα που έχουμε σήμερα. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα ακριβώ για να μπορούμε να επενδύσουμε. Ζητήσαμε επίσης και αύξηση των μισθών, κάτι το οποίο θα βοηθούσε μια οικονομία η οποία είναι διαρθρωτικά αποπληθωριστική. Θέλουμε επίσης καλύτερη ρύθμιση από πλευρά τη τράπεζα και των οικονομικών για να προστατεύσουμε καλύτερα τον Ευρωπαίο πολίτη. Εννοείται ότι είμαστε υπέρ ενό συντονισμού των δημοσίων πολιτικών, εννοείται και των οικονομικών πολιτικών, αλλά ε, το κοιτάμε επίση και ρεαλιστικά το θέμα, έτσι όπω έχουν σήμερα τα πράγματα. Δεν μπορούμε δηλαδή πια να πηγαίνουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται μία μεταρρύθμιση επί τη ουσία εκ βάθρων για να μπορέσει να λειτουργήσει ικανοποιητικά και να προσανατολίσει σωστά την οικονομική και κοινωνική μας πολιτική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λαλούκ. Ερχόμαστε στο δεύτερο γύρο τώρα από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ο κύριος Μιλάρ, Ουγγαρία πρώτα. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμοι συνάδελφοι, αξιότιμοι βουλευτές, ε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα για τη διαδικασία SPD που έχει δρομολογηθεί και όσον αφορά την Ουγγαρία υπάρχει αυτή η διαδικασία για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους ε, στόχους μας ε, σχετικά με το χρέος και το έλλειμμα. Προβλέπεται το 1% που πρέπει να δημιουργηθεί ως απόθεμα. Ε, τα βρίσκω σωστά αυτά που είπε η Επιτροπή, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αντέδρασε η Ουγγρική κυβέρνηση την ε, θέση της Ουγγρικής κυβέρνησης, την θεωρώ λαθασμένη, διότι τώρα στην Ουγγαρία η ανάπτυξη ανέρχεται σε 3 ή περίπου 4%. Ε, μάλιστα και πάνω από το 4% ήταν η ανάπτυξη ε, πέρυσι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η ε, ουγγρική οικονομία είναι υπερθερμασμένη και αυτό οφείλεται στο γεγονός ε, ότι ε, ανεκλήθησαν ταχύτατα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της ανάπτυξης των τομέα των κατασκευών κατά περίπου 50%. Και αυτό βέβαια ήταν μια φούσκα, φούσκα στον τομέα κατασκευών. Είναι ένα σαφές δείγμα της υπερθέρμανσης, αυξάνεται ο πληθωρισμός, ε, ε, το γκρικό νόμισμα ε, υποβαθμίζεται συνεχώς χάνει από την αξία του. Πέρυσι είχαμε γενικές εκλογές στην Ουγγαρία, φέτος έχουμε δημοτικές εκλογές. Ε, βλέπω λοιπόν να ελοχεύει ένας πολύ μεγάλος ε, κίνδυνος όσον αφορά αυτή την ε, τεχνητή ανάπτυξη, κατά την άποψή μου, όπως σας είπα, είναι μια φούσκα που θα σκάσει και γι' αυτό το λόγο εγώ χαιρετίζω τη σύσταση της Επιτροπής. Ε, ήπιος δανεισμός ε, είναι κάτι ε, το επιθυμητό και θα θέλαμε αυτή η φούσκα να περιστεί στο 2 μέχρι 3%. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κορογιάννης από την Ελλάδα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ ως πρόεδρος της ε, Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της ε, Βουλής των Ελλήνων χαιρετίζω τη σημερινή συνεδρίαση. Όπως γνωρίζετε η Ελλάδα από τον περασμένο Ιούλιο έχει μια νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η νέα κυβέρνηση έχει θέσει σε προτεραιότητα την ισχυρή ανάπτυξη με επενδύσεις, τους λιγότερους φόρους, την ποιοτική δημόσια υγεία και εκπαίδευση, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αναγέννηση του πρωτογενή τομέα, την αλληλεγγύη σε όσους έχουν ανάγκη, τη φύλαξη των συνόρων και την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σημειώσω ότι η Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωπη με κατακόρυφη αύξηση ροών μεταναστών μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ξεπέρασαν τους 2.500 οι μετανάστες που εισήλθαν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της έκθεσης για τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ, σημειώνουμε ότι οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στις δημοσιονομικές πολιτικές και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν. Στόχος μας είναι η αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ισορροπιών, η ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της ψήφισης ενός νέου αναπτυξιακού νόμου που κατατίθεται στη Βουλή τις επόμενες ημέρες και αφορά τις επενδύσεις του τομείς του τουρισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank uh, Ευχαριστούμε πολύ. Ευρωβουλευτής τώρα. Ο Λουί Καρικάνο από το Ρινιού, που είναι και σκιώδης εισηγητής. Αλλά κάθεται εκεί που κάθεται το ΕΛΚ κανονικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ όλους τους συνοδέρφους από τις άλλες χώρες που έχουν έρθει σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες. Στις διαπραγματεύσεις έδειξε η Renew ότι είμαστε ένας εταίρος που θέλει συμβιβασμούς και θέλει αναγέννηση της Ευρώπης πράγματι. Και ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια την κυρία Έστερ Ντελάνγκε. Εμείς θέλουμε να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις που πραγματικά χρειάζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είπαμε και χτες στον κύριο Ντράγκη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα νόμισμα που δεν χρειάζεται διάσωση, δεν χρειάζεται να το σώζει κανείς. Γι' αυτό και χώρες μέλη πρέπει να κάνουν ό,τι πρέπει, αλλά και οι νομοθέτες της χώρες μέλη πρέπει να κάνουν το δικό τους κομμάτι. Να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση, να υπάρχει η σταθροποιητική αυτή λειτουργία που θέλουμε, να υπάρχουν ε, ε, μεταρρυθμιστικά προγράμματα. Αυτά είναι προτεραιότητες που απαιτούνται για να αποφύγουμε να ξαναζήσουμε το 2012. Αλλά εδώ δεν πρόκειται μόνο για τη σταθερότητα της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεταρρυθμίσεις και ενόψη του μέλλοντος. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Πρέπει να έχουμε υγιή ε, δημοσιονομικά στις διάφορες χώρες και πρέπει και το νόμισμά μας να είναι ισχυρό, κατά το οποίο θέλουμε για τους πολίτες και για όλους. Και οι οικονομίες μας θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την ψηφιακή επανάσταση. Γι' αυτό και για μας ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι ζωτική σημασία. Και ελπίζω οι χώρες να υιοθετήσουν τις συστάσεις. Προς το παρόν 60% μόνο των συστάσεων έχουν υιοθετηθεί και ληφθεί υπόψη από τις χώρες μέλη, το οποίο δεν φτάνει. Εμείς δεν θα καθόμαστε να περιμένουμε σταυρωμένα τα χέρια ως Renew. Θέλουμε οι μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν. Η Ευρώπη λοιπόν έχει πολλά να κάνει. Και η υπόσχεση που δώσαμε για την αναγέννηση της Ευρώπης, εμείς θα την τηρήσουμε. Ευχαριστούμε. Τώρα, ο κύριος Φόρκη από την Ιταλία από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποια πράγματα έχουν αλλάξει στην Ιταλία από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ. Την περασμένη φορά ήμουν στην πλειοψηφία, τώρα είμαι στην αντιπολίτευση. Όμω ε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, Χωρί να γίνουν εκλογέ, συμβαίνουν στην Ιταλία. Αυτό όμω που δεν αλλάζει, κατά την άποψή μου, είναι το μεγάλο λάθος που βρίσκεται στη βάση των ε, ειδικών συστάσεων χώρα. Εγώ βασίζομαι στον πίνακα, στο scoreboard για την διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών και βλέπω ότι η Ιταλία ε, ουσιαστικά βρίσκεται εκτός παραμέτρου για το χρέος αυτό από την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και βέβαια έχουμε και ε, πολλούς ε, συντρόφους εδώ, 15 κράτη ακόμη και για την ανεργία. Καμία άλλη παράμετρος δεν είναι εκτός κλίμακας. Τώρα, για την ανεργία θέλουμε να τη μειώσουμε πώς. Με επενδύσεις και με μείωση της φορολογίας ή με πράγματα που προσπαθήσαμε να κάνουμε στο παρελθόν. Γιατί βλέπω εδώ τις ειδικές συστάσεις σαν χώρα και βλέπω ότι επί της ουσίας προτείνεται μείωση των δαπανών, αύξηση των φόρων και συγκεκριμένα ε, για τα νοικοκυριά και μείωση των συντάξεων. Αυτά τα έχουμε ήδη κάνει στην Ιταλία. Ήδη έγιναν από την κυβέρνηση Μόντι και ίσως κάποιος θα το θυμάται. Και έγιναν με βίαιο τρόπο γιατί είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση των φόρων στην νοικοκυριά, πολύ μεγάλη μείωση στη συντεξιδοτική δαπάνη, ο νόμος Φορνερό, όπως τον αποκαλούμε, και πολύ μεγάλο περιορισμό στις δαπάνες, περικοπές στις δαπάνες. Είχαμε 13 τετράμινα ύφεση, όχι μήνες, και οδηγηθήκαμε σε πολύ μεγάλη αύξηση της ανεργίας. Αν τώρα η μόνη παράμετρος που θέλουμε εδώ ε, βέβαια έχουμε και το θέμα του χρέους, γιατί η σχέση χρέους με το ΕΠ μετά από 13 τετράμινα ύφεση έχει χειροτερέψει, γιατί μειώθηκε το ΕΠ Τώρα, αν ε, ε, είμαστε μόνο εκτός σε δύο παραμέτρους, δηλαδή στο χρέος και στην ενεργεία σε σχέση με το scoreboard, πώς μπορείτε να συμβουλεύετε στην Ιταλία να ενεργοποιήσει πολιτικές που οδηγούν σε αύξηση του χρέους σε σχέση με το ΕΠ και αύξηση της ανεργίας. Ήδη τα έχουμε δοκιμάσει όλα αυτά. Γιατί μπορεί επί χάρτου είναι έτσι ε, να λέτε ότι θεωρία και πρέπει να τα δοκιμάσετε. Όχι, τα έχουμε δοκιμάσει όμως και να ακολουθήσουμε τις ίδιες ακριβώς συστάσεις μας λέτε που έγιναν άλλη στιγμή. Αν εμείς ήμασταν κυβέρνηση, τώρα είτε εμείς είμαστε κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, θα πρέπει να αντιταχτούμε σε αυτή την πολιτική και σε τέτοιο σύστημα και το είπε και ο Τράγκη. Ε, προχθέσαν, ε, δηλαδή ο Ντράγκη είναι το μοντέλο σας, ακόμη και αν λέει πράγματα που είναι κατά του δικού σας μοντέλου, θα πρέπει να τον ακούτε. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Ο κύριος ε, από τη Γερουσία, από την Ιταλική Γερουσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που μα καλέσατε να συμμετέχουμε σε αυτή τη συνεδρίαση. Μιλώ ω ε, γραμματέας ε, της Επιτροπής Προπολογισμού της Γερουσίας. Και είμαι πεπισμένο φιλευρωπαίος ε, και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και συνεργάζομαι με τους συναδέλφους στην Επιτροπή Προπολογισμού της Ένωσης. Είναι κρίμα που μόνο εννέα χώρες εκπροσωπούνται σήμερα. Ίσως θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα στο εγγύς μέλλον στην ε, ακρόαση του κυρίου Ντράγκη ακούσαμε ότι για μια ακόμη φορά έγινε εκτεταμένη χρήση κατά την άποψή μας ε, χρήσιμη των ε, εργαλείων της νομισματικής πολιτικής. Και θέλουμε τώρα να επισημάνουμε σε όλους τους συναδέλφους στο Κοινοβουλίο και στην Κομισιόν ότι πρέπει να επιμείνουμε επί των μέσων της δημοσιονομικής πολιτικής και οι δύο προτάσεις ε, που παρουσιάστηκαν. Η ε, μία που αφορά το σύστημα ε, για την προστασία των επενδύσεων, την προκυκλικότητα στις επενδύσεις ε, και το άλλο που αφορά το σύστημα ασφαλίσεων για να προστατευτούν οι δημόσιοι προπολογισμοί κατά τη διάρκεια των υφέσεων είναι ευπρόσδεκτες και θέλουμε να εργαστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους τομείς αυτούς. Uh, Ευχαριστούμε. Ο Έμες Ουρτασόν, ε, από τους Πρασίνους, που είναι επίσης και όδης εισηγητής Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ πολύ και εγώ καλωσορίζω θερμά εδώ τους φιλοξενούμενους μας σήμερα το απόγευμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο διάλογος αυτός είναι πολύ σημαντικός για να συντονίσουμε καλύτερα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε σχέση με το τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το οποίο χρειάζεται ε, βαθιά μεταρρύθμιση. Η δημοκρατική λογοδοσία, η ε, εξοικείωση του κόσμου με αυτό και ο ενστερνισμός του από πλευράς του κόσμου. Ε, χρειάζεται κάποια ενημέρωση επίσης για να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επικρίνει πολλές φορές ε, τα πράγματα για το βαθμολόγιο, για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπαμε πολλές φορές ότι ήταν πολύ αυστηρή και ήθελε να επιβάλλει τους δημοσιονομικούς κανόνες. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και άλλοι κανόνες που έχουν να κάνουν με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επέμεινε τόσο πολύ να τηρηθούν αυτοί οι κανόνες οι προκλήσει που έχουμε μπροστά μα είναι πολλέ. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, αναμφίβολα. Και σίγουρα πρέπει να συντονίσουμε τι οικονομικέ μα πολιτικέ. Αλλά με την έκθεση που έχουμε μπροστά μα τη κυρίας Δελάνγκε πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το εργαλείο αυτό, να κάνουμε κάποιε συστάσει για το πώ μπορεί αυτό να βελτιωθεί. Και ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι είναι σημαντικό, παλιότερα οι συστάσεις αυτές σαν χώρα δεν αναφέρονταν σχεδόν καθόλου στο θέμα της φορολόγησης, που είναι και αυτό σημαντικό. Και το άλλο που έχω να πω είναι ότι οι συζητήσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για να προβληματιστούμε γύρω από τον τρόπο με τον οποίο εκπονούνται οι οικονομικές πολιτικές. Και αυτό που χρειάζεται επίσης στην έκθεση είναι ότι το μείγμα πολιτικής που χρειαζόμασταν μέχρι τώρα, που έχει να κάνει κυρίως με τα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και το θέμα της ε, προσφοράς, όλα αυτά τελικά μάλλον κακό έκαναν στο περιβάλλον, αλλά και στην οικονομία δεν βοήθησαν. Οπότε η καθοδική πορεία που διαπιστώσαμε πρέπει να μας προβληματίσει. Και είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή. Όπως είπε και ο κύριος Δράγκη χτες, το δημοσιονομικό εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται. Υπάρχουν χώρες που έχουν περιθώρια, πλεονάσματα και που θα έπρεπε να τα χρησιμοποιήσουν επίσης. Συζητήσαμε και για τις διαφθορτικέ αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο, αλλά πρέπει να γίνουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαφθορτικέ μεταρρυθμίσεις. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έχουμε με την Ευρωζώνη είναι ότι δεν ολοκληρώθηκε αυτό που έπρεπε να ολοκληρωθεί και ξέρουμε ότι πρέπει μετά από την κρίση. Και είναι δηλαδή οι ασφαλίσεις καταθέσεων και η δημοσιονομική ικανότητα για να αντιμετωπίζουμε αντικυκλικές περιόδους. Οπότε ο διάλογος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σίγουρα βοηθάει πολύ με τα εθνικά κοινοβούλια. Ελπίζω η έκθεση αυτή, στην οποία συνεργαζόμαστε με την κυρία Ντελάνγκε, θα βοηθήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Για όσου ήρθαν αργά, υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να πάρετε το λόγο για να συμμετέχετε στη συζήτηση, πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το δελτίο, αυτό το χαρτί, το κίτρινο, και να το δώσετε σε κάποιο κλητήρα. Επόμενος γύρος τώρα. Ο κύριος Βίσσερα Λουξεμβούργο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας σήμερα το απόγευμα να είμαι εδώ. Θα αρχίσω υπογραμμίζοντας πόσο μεγάλη σημασία έχει η ανάλυση, δημοσιονομική ανάλυση που προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χώρες μέλη και κυρίως ε, για έναν βουλευτή από την αντιπολίτευση είναι πολύ σημαντικό να έχει ε, την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο. Τώρα για το Λουξεμβούργο και την οικονομική πολιτική και τις συστάσεις που γίνονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είμαστε στο πράσινο ως επιτοπλίστος στο Λουξεμβούργο. Έχουμε 20% δημόσιο χρέος και μια ανάπτυξη που είναι της τάξεως 2,5%. Δηλαδή, οι οικονομικοί δείκτες δεν είναι κακοί, δεν είναι αυτό το πρόβλημα στο Λουξεμβούργο, αλλά αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει στο Λουξεμβούργο είναι το μέλλον, το τι θα συναντήσουμε στο μέλλον. Αυτό πρέπει να απασχολήσει τη χώρα μου. Οπότε οι συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής πολύ σωστά υπογραμμίζουν τους μακροπρόθεσμους αυτούς κινδύνους για το Λουξεμβούργο. Πρώτα απ' όλα την βελτίωση της βιωσιμότητας ε, μακροπρόθεσμα του συνταξιδοτικού συστήματος. Για μας είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί το συνταξιδοτικό ε, σήμερα οδηγεί ακόμα σε θετικά αποτελέσματα, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε λίγα χρόνια, ήδη από το 2023 δηλαδή, θα έχουμε το αντίθετο. Και από τα μέσα ε, της δεκαετίας του 30 θα διάσουν τα ταμεία. Οπότε η σύσταση που γίνεται και που λέει ότι σήμερα ήδη πρέπει να καθορίσουμε ποιο θα είναι το σύστημα, ότι πρέπει να το αλλάξουμε, να το προσαρμόσουμε τώρα που είναι ακόμα καλά τα οικονομικά μας, είναι πολύ σημαντικό. Όντω έτσι πρέπει να γίνεται και πρέπει να τονίσουμε το ότι σήμερα πρέπει να γίνει αυτό. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αντικατοπτρίζεται πάρα πολύ καλά στις συστάσεις είναι ότι σήμερα γνωρίζουμε μία οικονομική εξέλιξη και μία οικονομική μεγένθηση ε, προφανή προς το 2,6-3% αλλά είναι δημογραφική και όχι παραγωγικότητας. Δηλαδή τα 10 τελευταία χρόνια αυξήθηκε ο πληθυσμός κάπου 20%. Και αυτό βέβαια έρχεται με διάφορα προβλήματα ότι αυξάνονται τα προβλήματα κατοικίας. Οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται κατά πολύ, 6-7%. Ε, οι δημόσιες μεταφορές ε, ξαφνικά βρίσκονται σε πρόβλημα γιατί φορτώνονται υπερβολικά. Οπότε οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς ε, που πρέπει να γίνουν είναι κάτι που γίνεται αισθητό καθημερινά. Η κυβέρνηση λοιπόν κάνει μεγάλες προσπάθειες. Σήμερα όμως τα προβλήματα δεν είναι τόσο προβλήματα χρηματοδότησης όσο προβλήματα εργατικού δυναμικού. Η ανάλυση λοιπόν που γίνεται είναι ορθή. Στο Λουξεμβούργο σήμερα πρέπει κυρίως να τονίσουμε την ε, εφαρμογή και την υλοποίηση των συστάσεων αυτών. Αυτό πρέπει να γίνει. Κύριος Πέσκο λοιπόν από την Ιταλία, από τη Γερουσία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω με πολλού Ευρωπαίου συναδέλφου που μιλάνε, που ασχολούνται με το ίδιο θέμα όπω και εμεί, με τον προπολογισμό. Ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί μα δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για του μακροοικονομικού δείκτε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το να αναλύει κανεί του δείκτε αυτού. Είναι δείκτε μακροοικονομικών ανισορροπιών που κατά την άποψή μα μπορούν να βελτιωθούν ε, μέσω δύο ο ένας παράγον είναι να μην υπάρχει ε, φορολογικό dumping. Αρκετές ε, χώρες ε, επ' αυτού προσπαθούν να ζημιώσουν άλλες χώρες, να προσφέρουν διαφορετικές δυνατότητες. Και δεύτερον, ε, όσον αφορά την εργασία. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλέ διαφορές. Ε. Μην ξεχνάμε ότι πολλές εταιρείε ε, μετακομίζουν σε άλλες χώρες γιατί εκεί βρίσκουν καλύτερες ρυθμίσεις. Άρα δηλαδή αυτοί οι μακροοικονομικοί δείκτες μπορούν να ληφθούν υπόψη και με τον τρόπο αυτό να κατανοήσει κανείς καλύτερα το τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες. Αυτό που θα ήταν χρήσιμο πλευράς μεθόδου είναι να συσταθεί ένας και μόνος δείκτης ε, που θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους άλλους δείκτες που συζητάμε εδώ. Όχι με την έννοια της ταξινόμησης, ε, αλλά με την έννοια ενός δείκτη που θα παρουσιάζει και τη θέση κάθε χώρας έναντι των υπολείπων. Αυτά όσον αφορά τη μέθοδο. Όσον αφορά όμως τα θέματα πολιτικής εφήσεως, ε, πολιτικής οικονομίας, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο ε, να ε, εξετάσουμε όλοι μαζί προβλήματα που αφορούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αναφέρομαι στους νέους, στην τεχνολογία, στην παιδεία, στην υγεία, στο περιβάλλον, ε, στο θέμα της ε, τρίτης ηλικία. Αναφέρθηκε προηγουμένως, ε, όλοι κάτι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά αυτό το θέμα, γιατί αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας. Και τέλος, να ασχοληθούμε με την εργασία. Σε όλους αυτούς τους τομείς πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Δυστυχώς όμως ε, πολλές χώρες δεν έχουν ε, πολλές δυνατότητες γιατί ε, γνωρίζουμε ότι έχουν περικοπεί τα κονδύλια. Κατόπιν τούτου θα ήθελα να σας παρακαλέσω ή μάλλον απευθύνω έκκληση σε όλες τις χώρες όπως συμβαίνει, όπως ανέφερε και η νέα επίτροπος, η κυρία Λάιν, το ότι θα υπάρξει μια νέα συμφωνία για το περιβάλλον, να δούμε πού ε, είναι αυτοί οι τομείς όπου μπορούν να γίνουν επενδύσεις ε, που να διαφοροποιούνται από τους κανόνες του προπλογισμού, γιατί υπάρχουν κανόνες του που απαγορεύουν σε ορισμένες χώρες να προβούν σε επενδύσεις. Πολύ ωραία. Πάω τώρα στον κατάλογο των μελών του Κοινοβουλίου από το ECI. Άρ, που είναι και ο Δεν έχουμε κανένα από, τους, ε, από την ομάδα ID, γι' αυτό πάω πάλι στο ECR. Ευχαριστώ κύριε Μάιερ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της και νομίζω λέει ο κύριος Γιουρτσίκα ότι μας παρουσίασε μια πολύ καλή έκθεση και εκτιμώ ε, και τις προσπάθειες που έχει καταβάλει στις ε, ε, συναντήσεις των σκιωδών να καταθέσει ένα ισορροπημένο κείμενο. Ήδη είχαμε δύο συνεδριάσεις και θα υπάρξουν άλλες δύο με τους σκιώδεις, όμως πρέπει να σας πω ότι έχω απογοητευτεί λιγάκι όσον αφορά την ενσωμάτωση των τροπολογιών από ορισμένε πολιτικές ομάδες. Το κείμενο τώρα είναι πολύ χειρότερο και βεβαίως ορισμένες χώρες ενδεχομένως να μην θέλουν ε, τη λύση της αγοράς για να λυθούν τα προβλήματα του ευρώ. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι διαγράφεται, ε, διαγράφονται και σημαντικές ε, παραπομπές σε γεγονότα ε, παραδείγματος χάρη να μην αναφέρεται το προφανές στην παράγραφο 13 ότι οι δημόσιες επενδύσεις κυρίως ε, χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους. Δεύτερον, το κείμενο ε, γίνεται πολύ πιο ήπιο εκεί που γίνεται λόγος για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που αναφέρεται ότι δεν πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως το σύμφωνο αυτό. Εμάς δεν μας αρέσουν αυτά, ε, γιατί όταν μιλάμε ε, δημόσια, μιλάμε συνεχώς για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, για φορολογία, αλλά κατά κάποιον τρόπο όταν φτάνουμε στους κανόνες που διέπουν τους δημόσιους θεσμούς, εκεί ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή η αντίδραση είναι υπεύθυνη. Και θέλω να πω ότι υπάρχουν ε, και κάποιες ε, τροπολογίες συμβαστικές ε, που δεν μπορώ να δεχτώ, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι τα φορολογικά θέματα καλύτερα να παραμείνουν στα χέρια των κρατών μελών και οποιαδήποτε κοινή αντιμετώπιση θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο. Έχουμε και άλλο ένα αίτημα από μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου, κύριο Σατήλα, από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Ούγγρος συνάδελφος που πήρε το λόγο προηγουμένως βρίσκεται στα έδρανα της αντιπολίτευσης και είπε τα ίδια επιχειρήματα τα, με τα οποία συγκρουστήκαμε όταν εγκρίναμε τον προϋπολογισμό. Μπορώ να πω ότι είναι κάπως λανθασμένα τα συμπεράσματα. Εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερα να επιστρέψουμε στο σχέδιο, στο νομοσχέδιο που εξετάζουμε. Σύμφωνα με την πρόταση της Ουγγαρίας, η διαδικασία που έχει ξεκινήσει κατά της Ουγγαρίας μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά ζημιών στην εγκαρία. Θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει μια σειρά ζημιών. Και θα αναφερθούν σύντομα από τον Υπουργό τα μέτρα που θα ληφθούν. Σε ό,τι αφορά τις ειδικές συστάσεις αναχώρα, Έχουμε διάφορες ε, προτάσεις ε, για την ε, βελτίωση του συστήματος υγείας και άλλα δημοσιονομικά μέτρα. Αλλά σε ό,τι αφορά τα μέτρα που προτείνονται σε φορολογικό επίπεδο, εμείς δεν συμφωνούμε. Και σε ό,τι αφορά το έλλειμμα, πρέπει να έχουμε κατά νου το αποτέλεσμα που θα επιφέρουν τα μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος. Εμείς είμαστε υπέρ της βιωσιμότητας στη διαχείριση του προϋπολογισμού και την αποδοτικότητα των δαπανών. Εδώ και μήνες γίνεται αναφορά στη συζήτηση για τους τρόπους επικαιροποίησης των δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό τα δεδομένα να επικοινωνούνται σωστά. Επίσης, ε, είναι πολύ σημαντικό και το θέμα του ενστερνισμού των μέτρων από την πλευρά των κρατών, το ownership. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνα θα πρέπει να ξεκινήσει ένας ε, διάλογος σε ό,τι αφορά παραδείγματο χάρη κάποιε συστάσει ε, που έχουν διατυπωθεί στον τομέα τη γειτοσύνη αφορούν περισσότερο ε, την πολιτική παρά το θέμα του προπολογισμού και για μας αυτό δεν είναι αποδεκτό. Ευχαριστούμε κυρία Τίλα. Δεν βλέπω να ζητά κάποιο άλλο το λόγο από τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε το λόγο, γιατί έχουμε χρόνο στη διάθεσή μα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Γκουσμά από την ΚΟΕ, που είναι επίση σκιώδη εισηγητή στην έκθεση τη κυρία Ντελάνγκε. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες ε, έχουν ε, αποκαλύψει μια προκυκλικότητα, όπως αποκαλείται. Στην έκθεση αυτή προσπαθούμε να εισαγάγουμε κάποιες ε, ιδέες που παραπέμπουν στη δημιουργία εργαλείων που να ε, μειώνουν ε, αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, είτε τη δημιουργία μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα προσανατολίζονται στις επενδύσεις και στις επενδύσεις σε τομεί που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές πολιτικές και στην απάντηση στην κλιματική αλλαγή. Εμείς ε, θα θέλαμε επίσης να εισαχθούν κάποιες εξαιρεσει στην εφαρμογή των κανόνων του Σύμφωνου σταθερότητα και Ανάπτυξης που να επικεντρώνονται στι επενδύσει σε αυτούς τους τομείς. Και ε, αυτό ε, μπορεί να συνάδει με ορθούς δημοσιονομικούς ε, κανόνες που να έχουν μία αντικυκλική πολιτική. Και τώρα θα ήθελα να δούμε πώς πρακτικά μπορούν να ε, υλοποιηθούν κάποιες διακηρύξεις που όπως πρέπει το χάρη είναι πολέμηση της στόχης και της κλιματικής αλλαγής. Αν αυτές οι προτεραιότητες, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα αντιμετωπίσουν σοβαρά, τότε θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται όλα αυτά και θα πρέπει να έχουν συνέπειες στο πώς ε, κατανοούμε τους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, εδώ, σε σχέση με τη συζήτηση για τις ειδικές συστάσεις αναχώρα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδες να κάνουμε έναν ε, ε, κριτικό απολογισμό. Δηλαδή, έχουμε πολλές δημοκρατικές χώρες που νόμιμα ε, επιλέγουν να μην ακολουθήσουν αυτές τις συστάσεις, γιατί δεν συνάδουν με το πρόγραμμά τους. Αλλά επίσης να αξιολογήσουμε και τι έγινε με τις χώρες που ακολούθησαν τις συστάσεις αυτές. το χάρη, μπορεί να έχουμε μία πολύ λίγο συγκεκριμένη σύσταση που μπορεί να εφαρμοστεί εφαρμοστεί σε όλες ε, τις χώρες, παραδείγματο χάρη να υπάρχει ευελιξία στην αγορά εργασία. και μπορεί να οδηγήσει ε, τις χώρες ε, στο να καταργήσουν συλλογικές συμβάσεις με την υπόσχεση ότι θα έχουμε μεγαλύτερη απασχόληση και ψηλότερους μισθούς. Και αυτό δεν υλοποιήθηκε και ε, βλέπουμε διάφορες γενιές που έχουν επηρεαστεί από αυτές εργασιακές μεταρρυθμίσεις. Άνθρωποι θίγονται από πιο χαμηλούς ε, μισθούς και από την επισφάλεια παρόλο που έχουν υψηλά προσόντα. Αυτά τα θέματα εμείς ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει, σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να δοθεί απάντηση. Επίσης, θεωρούμε ότι στο θέμα των μακροοικονομικών ανισορροπιών, επί το οποίο δημιουργήθηκε μία σειρά δικτών, θα πρέπει επίσης να εκφράζεται στις ευρωπαϊκές πολιτικές, γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα ουσιαστικά είναι ότι έχουμε γραφειοκρατικές συστάσεις χωρίς να γίνεται τίποτα στις ευρωπαϊκές πολιτικές και πολύ λιγότερο στις εθνικές πολιτικές. Thank you uh, Σας ευχαριστούμε. Τώρα, συζήτηση μεταξύ μας. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει το λόγο, εφόσον έχει συμπληρώσει βέβαια το κίτρινο χαρτί. Λοιπόν, οποιοδήποτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια ή άλλος θέλει το λόγο, παρακαλώ. Έχω ήδη τον Ερκαγκέρικα από το ΕΛΚ πάντως εδώ στον καταλογό μου που έχει συμπληρώσει το κίτρινο χαρτί. Ευχαριστώ, ναι, κύριε και εγώ χαιρετίζω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η σύνθεση που μπορούμε δηλαδή μεταξύ μας να συζητάμε ε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμενο με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα περισσότερα από αυτά τα θέματα είναι είτε ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, είτε εθνική αρμοδιότητα, είτε μεικτή. Τώρα θα μιλήσω ουγγρικά. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία το να ακούσουν οι συνάδελφοι και όχι μία, δύο-τρεις φορές την πολύ ωραία ουγγρική μας γλώσσα. Ε, τώρα, όσον αφορά το εξάμεινο, ε, θέλω να σας πω ότι το θέμα δεν είναι να ε, μεταφέρουμε εδώ εσωτερικοπολιτικές συζητήσεις. Μιλώντας για την Ουγγαρία και συγκρίνοντας ε, την κατάσταση ε, τότε ε, πριν από 10 χρόνια όταν η Ουγγαρία για πρώτη φορά έπρεπε να διασωθεί, σήμερα μην ξεχνάμε ότι έχουμε ανάπτυξη της τάξης του 5%, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 5 χρόνια το θέμα της ε, απασχόλησης. Από το 56% φτάσαμε στο 70%. Ε, το χρέος ε, μειώθηκε σε κάτω από 70%, ήταν παλαιότερα πάνω από 80%. Αυτούς τους δείκτες δεν μπορεί κανείς να τους αμφισβητήσει. Το εξάμεινο είναι ένα θαυμάσιο οικονομικό εργαλείο αλλά θα πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι αν θέλουμε τελικά να τα βάλουμε όλα σε αυτό το εξάμεινο, τότε θα χάσουμε πολύ περισσότερα από το να ε, χρησιμοποιήσουμε αυτό το χρήσιμο εργαλείο αποτελεσματικότερα. Γιατί τελικά ε, υπάρχει κίνδυνος ε, να έχουμε ένα πολυφορτωμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και το εξάμεινο είναι ένα πολυφορτωμένο δέντρο. Η Κομισιόν προσπαθεί τώρα να ε, χαρακτηρίσει κάτι ως εξάμεινο που δεν έχει όμως καμία σχέση με τον πολιτικό συντονισμό. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι χώρες ε, θα έχουν την αίσθηση ότι δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Ακούσαμε το θέμα της ε, ιδιοκτησίας, της οικειοποίησης είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτό ειδικά ε, θα χαθεί εάν ε, τελικά το εξάμεινο δεν ερμηνευτεί σωστά. Στα αγγλικά τώρα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που αφορούν περισσότερο στην εναρμόνιση των φόρων και προβλέπουν ε, την ψηφοφορία με ειδική ε, πλειοψηφία ή καθορίζουν ελάχιστα ε, ποσοστά χρέους. Ο συνάδελφος μόλις βγήκε από το ECR είπε κατ' ουσίαν ότι προβολούμε μόνοι μας το πόντι μας. Γιατί διότι αν δεν επιτρέψουμε τον φορολογικό ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα φύγουν εταιρείε. Εγώ πιστεύω ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι καλός γενικότερα για τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό εγώ είμαι υπέρ αυτών των τροπολογιών που προβλέπουν την φορολογική εναρμόνιση. Ευχαριστούμε τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Μπέλκα. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει δύο προβλήματα. Το ένα είναι η χαμηλή ανάπτυξη και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την ανταγωνιστικότητά μας διεθνώς και το δεύτερο πρόβλημα είναι η απόκληση. Ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τη συνοχή με το ίδιο το μέλλον της Ευρωζώνης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Κάποιες χώρες αναπτύσσονται πιο γρήγορα από άλλες, κάποιες έχουν χαμηλότερο πληθωρισμό από άλλες. Αυτό είναι ένα γεγονός. Μέσα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε σημαντικά εργαλεία όπως είναι εκείνο για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δεν ξέρω κατά πόσο το χρησιμοποιούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το χρησιμοποιεί, δεν ξέρω πόσο καλά. Αρκετά επιθετικά θα έλεγα και με συμμετρικό τρόπο. Δηλαδή δεν αφορά μόνο τις χώρες που έχουν μείνει πίσω, που πρέπει να αλλάξουν τις πολιτικές τους, αλλά ακόμα και αυτές οι οποίες πηγαίνουν υπερβολικά γρήγορα. Εγώ αυτό πιστεύω. Και λυπάμαι που σας το λέω, λέω έτσι είναι. Γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με το μέλλον. Έχουν να κάνουν με την ίδια την επιβίωση της Ευρωζώνης και του ευρώ. Ακούσαμε ότι δεν έχουμε αρκετές επενδύσεις στην Ευρώπη. Μα παντού ισχύει το ίδιο. Παντού και στις προηγμένες χώρες. Δεν ξέρουμε γιατί, άλλο ιδιωτικό τομέα δεν είναι πρόθυμος να επενδύσει σήμερα. Και είτε το θέλουμε, είτε όχι, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, ε, πρέπει να επενδύσει το δημόσιο. Πρέπει όταν βέβαια είναι αυτό εφικτό και όταν χρειάζεται, να έχουμε πιο εντατικά δημόσιες επενδύσεις. Αν έχετε κάποιες αφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των δημοσίων επενδύσεων επειδή είσαστε φιλελεύθερος, μα δεν έχουμε άλλη λύση, αφού δεν υπάρχουν επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε να πούμε στις χώρες, να πούμε στις κυβερνήσεις και αυτή είναι η έκκληση που κάνουμε και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντικαταστήσει τις ιδιωτικές, να τι συμπληρώσει, εν πάση περιπτώσει, από δημόσιες επενδύσεις. Ευχαριστούμε, Μάρκ. Να σα πω ότι έναν έχω ακόμα στον κατάλογο μου, οπότε αν κάποιο άλλος θέλει να συμμετάσχει στη συζήτηση, παρακαλώ να συμπληρώσετε το κίτρινο χαρτί. Εντάξει, εσά σας βλέπω, σα ξέρω. Αλλά αλλιώ καλό είναι να έχουμε το κίτρινο χαρτί, αλλιώ θα ολοκληρώσουμε. Η Ρομπέρτα Ρούλαντ έχει τώρα το λόγο. Μη, ο Ρόμπερτο Ρούλαντ, μη εγγεγραμμένο. Ευχαριστώ. Είναι τιμή για μένα που μπορώ εδώ να συμμετέχω στη συζήτηση αυτή. Άκουσα την συζήτηση, ήμουνα στις επενδυτικές αγορές για 30 χρόνια και παρακολουθώ κάθε χρόνο την ε, οικονομική πολιτική. Για μένα δύο είναι τα προβλήματα. Ένα είναι η χαμηλή ανάπτυξη και τι το προκαλεί αυτό το πρόβλημα και υπάρχει και το άλλο πρόβλημα όταν προσπαθείς να δημιουργήσεις ένα στενό κορσέ μια νομισματική πολιτική για 27 ε, χώρες. Ακούσαμε πολλά για τις δυσκολίες της Ευρωζώνης εξαιτία ε, εμπορικών εντάσσεων, εξωγενών παραγόντων κλπ. Αλλά δείτε στις Ηνωμένε Πολιτείες έχει ανάπτυξη 3% δημιουργία απασχόλησης, παραγωγικότητα σε επίπεδα που εμείς τα είχαμε τη δεκαετία του 80. Αν δείτε τα χθεσινά στοιχεία από την Γερμανία, από το Services PMI, τώρα μπαίνουμε σε αρνητικά επίπεδα. Έχουμε και μια υπαρξιακή κρίση η οποία αναδύεται στην Ευρώπη. Και το ζήτημα είναι πώς το λύνουμε αυτό. Κατά τη γνώμη μου, η λύση δεν είναι να κάνουμε αυτά που κάνει ιστορικά ο Ντράγκη, δηλαδή την ποσοτική χαλάρωση μαζικά, γιατί δημιουργεί ε, σοβαρά προβλήματα ε, με την κίνηση του κεφαλαίου, δημιουργεί τεράστια κόστη, χάνεται χρήμα. Οπότε η Ευρώπη σήμερα δεν έχει κανονικό κόστος κεφαλαίου. Οπότε αν ψάχνετε γιατί δεν υπάρχουν ιδιωτικέ επενδύσεις, γι' αυτό. Γιατί δεν δανείζουν οι τράπεζε στι επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν γιατί γνωρίζουν ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξη όπου δεν υπάρχει τελικά ε, πραγματικό κόστο κεφαλαίου. Οπότε τελικά όταν έχουμε πληθωρισμό σε μη παραγωγικό ενεργητικό, προφανώς θα καταλήξουμε σε φούσκα. Η λύση μου λοιπόν για την Ευρώπη είναι να αποφύγουμε αυτήν την κεντρική ιδέα ότι μπορούμε να δίνουμε ε, κεφάλαιο μέσα από αυτές τις νέες πράσινες ε, πολιτικές όπου το κράτος αποφασίζει που θα πάνε τα χρήματα. Είναι σφάλμα αυτό. Δείτε στη Γερμανία τι έγινε χτες. Προσπάθησε να εκδώσει ε, το ομόλογα του χρέους, όμως χωρίς την ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρχει λύση. Χρειάζεται απορρίθμιση, χαμηλή φορολόγηση και ενίσχυση της ιδιωτικής αγοράς. Δεν ζούμε σε μια οικονομία κεντρικά σχεδιασμένη, αλλιώς θα καταλήξετε σε μιζέρια. Ο κύριος Κίρτσος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, καταρχήν καλωσορίζω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια γιατί με τις παρεμβάσεις τους εμπλουτίζουν τον προβληματισμό μας ε, μας δίνουν να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στις χώρες τους και πώς ε, πρέπει να συντονιστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, θα σας πω ευθέως ότι δεν έχω τις λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ε, αλλά ακριβώς επειδή δεν έχω τις λύσεις, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε δημιουργική σκέψη. Αυτό σημαίνει ότι τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας πρέπει να τα αξιοποιήσουμε με σωστό τρόπο, αλλά πρέπει με διάφορους τρόπους να συμφωνήσουμε να πάμε και λίγο πιο πέρα, χωρίς πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά για να λύσουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Νομίζω ότι είμαστε σε μία περίοδο μεγάλης αστάθειας, ε, η οποία βέβαια μπορεί να εξελιχθεί θετικά ή αρνητικά. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι τα αρνητικά επιτόκια, ε, τα οποία είναι εντυπωσιακά. Δηλαδή καταλαβαίνω τον προβληματισμό πολλών συναδέλφων, ιδιαίτερα για παράδειγμα από τη Γερμανία. Από την άλλη τα αρνητικά επιτόκια ίσως είναι ένα αναγκαίο κακό σε αυτή τη φάση, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς να διαχειριστούμε την οικονομία. Μετά βλέπουμε μία έλλειψη οικονομικής δυναμικής, ε, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι οι πιο, οι πιο δυναμικοί χάνουν τη δυναμική τους. Ε, δηλαδή, ε, για παράδειγμα, πάλι η Γερμανία, επειδή είναι παγκοσμιοποιημένη η οικονομία της, πληρώνει ακριβότερα ε, από ότι, για παράδειγμα, μια οικονομία σαν την Ελλάδα, που είναι λιγότερο ενταγμένη στο διεθνές σύστημα, την, θα έλεγα, εμπορική κόντρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Επομένως πρέπει να τα δούμε και αυτά. Ε, είμαστε όλοι σε γενικές γραμμές υπέρ της πράσινης μετάβασης και του Green Deal, αλλά δεν ξέρουμε πώς ακριβώς να το εφαρμόσουμε, ώστε να τραβήξουμε πρόσθετες επενδύσεις ε, και να πάει καλύτερα η οικονομία. Παρακολουθούμε όλοι τον Brexit και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει, ούτε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ξέρουν. Ε, η δικαιοσύνη έχει στραφεί κατά τη κυβέρνηση, η κυβέρνηση κατά της δικαιοσύνης, ε, η κυβέρνηση κατά των κομμάτων, τα κόμματα κατά τη κυβέρνηση, Θα δούμε τι ακριβώ θα συμβεί. Ε, και έχουμε και ένα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Αναφέρθηκα πριν στα προβλήματα τα εμπορικά μεταξύ των ΗΠΑ και τη Κίνα. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, καμιά φορά και με αγωνία, τι γίνεται στη Σαουδική Αραβία και την ευρύτερη περιοχή. Άρα, το συμπέρασμα που βγάζω εγώ είναι ότι ε, έχουμε μια προκλήση να αντιμετωπίσουμε, όσο, όσο καλύτερα αξιοποιήσουμε τους κανόνες που έχουμε και όσο πιο δημιουργική σκέψη έχουμε όλοι μαζί, τόσο καλύτερα θα πάμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. So we have uh, uh, another members that uh, want to. Σας ευχαριστώ. Έχουμε και άλλα μέλη. κυρία Ντονάτο από το ID καταρχήν είχε ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα μιλήσω τελικά. Και εγώ υπό το φως ε, όσων ε, ακούστηκαν ε, και βάσει τον όσο είπε ο θα ήθελα να θέσω κάποιους προβληματισμούς για την οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για όλα τα θέματα που συζητούμε. Κατά την άποψή μου, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη σκοπιά της ανάπτυξης, Έχουμε δύο περιοχές με διαφορ... δύο ζώνες, δύο περιοχές που έχουμε διαφορετική εξέλιξη. Την Ευρωζώνη αλλά και τις χώρες που δεν ανήκουν στο ευρώ. Και από τα στοιχεία που έχουμε δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Τα τελευταία χρόνια κυρίως οι χώρε που βρίσκονται εκτό Ευρωζώνης έχουν αναπτυχθεί, ενώ οι χώρες της ευρωζώνη βίωσαν ε, είτε μία πολύ μικρή ανάπτυξη είτε μία περίοδο τελμάτωσης και ε, βέβαια είχαμε και κάποιες που αναπτύχθηκαν όπως η Γερμανία και τελικά σε αυτό το τέλμα εμπλέκονται όλοι. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε ε, επί της αποτελεσματικότητας και την ε, επικαιροποίηση των κανόνων που διέπουν την Ευρωζώνη. Μιλώ κυρίως ε, για ε, δεσμούς που αφορούν τον προϋπολογισμό. Αναφέρονται σε αυτά κυρίως οι ειδικές συστάσεις αναχώρας. Αναχώρα, με συγχωρείτε. Όπως είπε και ο πρόεδρος Τράγκη χθες, η αναγκαιότητα να αναθεωρηθούν αυτοί οι δεσμοί με το σύστημα υπό το φως ότι σήμερα φαίνεται να μην είναι πλέον αποτελεσματική, για να ε, μπορέσουμε να έχουμε αντικυκλικές πολιτικές για να ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο είναι μια πτυχή που όλοι θα πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη. Επίσης και σε ό,τι αφορά τις συστάσεις για χώρες όπως η Ιταλία να υλοποιήσει τις διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις πέρα από τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη δικαιοσύνη, τη μείωση της γραφειοκρατίας από τα οποίο δεν υπάρχει φυσικά εξαίρεση. Αλλά εμεί ω Ιταλία αλλά και η Ελλάδα έχουμε υλοποιήσει πολλέ από τις μεταρρυθμίσει που μα ζητήθηκαν. Και μιλώ για τη μεταρρυθμίση της αγορά εργασία, του τεξιδοτικού συστήματος. Έχουμε σεβαστεί τους ε, κανόνες τη τραπεζική εποπτεία. Όμως παρόλα αυτά δεν αναπτυσσόμαστε. Και αυτό που ζήτησε χτες ο πρόεδρος Τράκη, δηλαδή τα κράτη-μέλη που έχουν περισσότερο περιθώριο δαπανών να ασχοληθούν με την τόνωση της ανάπτυξης, επενδύοντας οι ίδιες και κάνοντας τις απαραίτητες δαπάνες σε αντικυκλικά πλαίσια, στην πραγματικότητα δύσκολα θα γίνει. Αυτή η έκκληση δύσκολα θα υλοποιηθεί, γιατί αν δεν υπάρχουν κυρώσεις και αν η προσέγγιση ε, πάντοτε φοβάται την αύξηση του πληθωρισμού, είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία, δεν θα αναλυφθεί αυτή η πρωτοβουλία που θα ωφελήσει όλες τις χώρες της Ευρωζώνης από την πλευρά των χωρών που θα μπορούσαν να το κάνουν, που είναι σε θέση να το κάνουν. Εν μεταξύ, χώρες ε, που θα μπορούσαν να δαπανίσουν ε, περισσότερο και που θα χρειάζονταν ε, ε, περισσότερες παρεμβάσεις σε διαρθρωτικό επίπεδο, σε υποδομές, στην παιδεία, αλλά και σε άλλους σημαντικούς τομείς για την ζωή των πολιτών, δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί τους, ζητού, τους ζητείτε να διατηρήσουν δημοσιονομικές πολιτικές πολύ προσεκτικές. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι ε, δεν μας οδηγεί πουθενά το να προσεγγίσουμε την κατάσταση με τον τρόπο αυτό. Όλοι θα πρέπει να το αναλογιστούμε αυτό. Γιατί απουσία μιας διεξόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, όπως αυτό που είπε ο Πρόεδρος, το να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα ε, προπολογισμού όπου μία νέα κεντρική αρχή θα αποφασίζει για όλους ε, πού θα γίνουν οι δαπάνες, πώς θα επενδύσουμε κτλ. Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι τα κρατημέλη διατεθειμένα να δεκτούν κάτι τέτοιο, σχεδόν ομόφωνα. Απουσία λοιπόν αυτού θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο η κρίση αυτή να ξεπεραστεί. Αν αφαιθούμε μόνο στην ελεύθερη πρωτοβουλία χωρών που έχουν μεγαλύτερο πλεόνασμα, αν αφαιθούμε λοιπόν στη δική τους βουλή να αυτές οι πολιτικές. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και επί ενός συστήματος κινήτρων αν όχι για τις χώρες αυτές, έχοντας και κατά νου την ύπαρξη ενός συνδέσμου για το πλεόνασμα, μέχρι τώρα δεν φαίνεται να έχει γίνει σεβαστό, ούτε μάλιστα έχουν επιβληθεί και κυρώσει. πόσο μάλλον δεν έχουν επιβληθεί κυρώσει. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Πέντρο από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε εγώ θα μιλήσω πορτογαλικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να συζητήσουμε περισσότερο και θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποια σχόλια των προλησόντων που με έκαναν και εμένα να πάρω το λόγο. Πράγματι, μιλάμε εδώ για την δημόσια οικονομική πολιτική και ήθελα να πω ότι ε, δεν θα μπορούσα παρά να διαφωνήσω με την ιδέα ότι η συνταγή θα ήταν να μην κάνουμε τίποτα, να απορριθμίσουμε και να αυξήσουμε τα επιτόκια και με ένα μαγικό τρόπο θα επιστρέψει η οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι το μοντέλο που το επερασπίζουν εδώ από την γιγάντια οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε, ακριβώς γιατί είχαμε ένα εντελώς απορριθμισμένο μοντέλο, ένα ε, μοντέλο το οποίο οδήγησε σε μακροοικονομικές ανισορροπίες διαφορετικές σε όλη την Ευρωζώνη και μάλιστα χρειάστηκε και η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να σώσει το ευρώ. Και τώρα φαίνεται σαν να συζητάμε εδώ μία άλλη πραγματικότητα. Από την άποψή μου, κατά την άποψή μου, εμείς χρειαζόμαστε ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον για να αντιμετωπίσουμε όλες τις οικονομικές συνέπειες είτε του Brexit, είτε της ε, σημερινής κατάστασης, είτε του εμπορικού πολέμου. Και γι' αυτό θα πρέπει οι χώρες με μακροοικονομικό πλεόνασμα να κάνουν περισσότερα και η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών να ενεργοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε κάποια θετικά σημάδια από τις χώρες αυτές, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη αποτελεσματικότητα. Χρειαζόμαστε τα εργαλεία σταθερότητα τη Ευρωζώνη που δεν τα έχουμε ακόμα, δηλαδή την δημοσιονομική ικανότητα τη Ευρωζώνη ε, και να υλοποιηθεί περαιτέρω η Τραπεζική Ένωση, προκειμένου η Ευρωζώνη να μπορεί να αντιμετωπίσει τα μελλοντικά σύμμετρα σοκ που θα λάβουν χώρα και συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε να δράσουμε από την ε, σκοπιά κάποιων παραγόντων που αφορούν την προσφορά. Ε, δηλαδή να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα ως προς το δημογραφικό αλλά και ποια θα είναι η δική μας ικανότητα να είμαστε καινοτόμοι. Θα ήθελα να φέρω και ένα άλλο στοιχείο στη συζήτηση, όμως ε, δεν πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την κούρσα προς τα κάτω σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Ακόμη και κάποιες χώρες που υλοποίησαν αυτό τον δημοσιονομικό ανταγωνισμό. Είδαμε ότι είχαν αρνητικές συνέπειε. εμείς αν συνεχίσουμε τον προηγούμενο δρόμο της, ε, του φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών θα εξαντλούσαμε την ικανότητά μας ε, να, να χρηματοδοτήσουμε το κοινωνικό κράτος και τις δημόσιες πολιτικές και τελικά θα περιορίζαμε πάρα πολύ την ικανότητά μας να αναπτύξουμε με βιώσιμο τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, ε, ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται προκλητική η δική μου παρέμβαση, όμως ε, θα ήθελα να συνεισφέρω στη συζήτηση που υλοποιούμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Εκ μέρους της συσχήτριά μας, επιτρέψτε μου όχι τόσο να συνοψίσω, όσο να κάνω κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις πριν ολοκληρώσουμε. Πρώτα απ' όλα, Υπόθηκε πολλές φορές μέχρι τώρα ότι η αρμοδιότητα της δημοσιονομικής πολιτικής είναι στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων. Όμως, στο ίδιο πλοίο βρισκόμαστε όλοι. Οι ευπάθειες, η κατάρρευση, η οικονομική κρίση του διπλανού μου θα οδηγήσει και εμένα στην πτώση. Οπότε, ε, χρειαζόμαστε ισχυρές οικονομίες παντού. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Είναι προς το συμφέρον όλων μας να είναι όλες οι οικονομίες καλά. Δεύτερον, πολλά υπόθηκαν για τις συστάσεις. Αυτό το οποίο είναι επίσης σημαντικό είναι ο ενστερνισμός. Ότι δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι το ωφέλει από την υλοποίηση των ε, συστάσεων είναι ωφέλη για τον ίδιο τον κόσμο. Τώρα, τα Εθνικά Κοινοβούλια έδειξαν πόσο πολύ τα ενδιαφέρει η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και η αναχώραση στάσης και μερικοί από εσά είπατε ότι θεωρείτε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην εσωτερική σα πολιτική. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Και από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντάξει, η συζήτηση είναι πολιτική, υπάρχει διάσταση απόψεων όσον αφορά τι προτεραιότητε. Δεν είναι η πρώτη συζήτηση, ούτε η τελευταία που κάνουμε. Θα συνεχίσουμε και σίγουρα και με τι συναντήσει των σκιωδών. Και στο τέλο ε, θα υπάρξει μια, πιστεύω, καλά ισορροπημένη έκθεση. Συνεπώς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους προσκεκλημένους μας πρώτα απ' όλα, αλλά και όλους όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ και όλους εσάς που παρακολουθήσατε τη συζήτηση. Όσον αφορά την οργάνωση, να ξέρετε 2 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή και στην Ολομέλεια επίσης τον Οκτώβριο πριν από τη συνεδρίαση την αντίστοιχη του Συμβουλίου. Το επόμενο θέμα μας είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Τίγκεσεν, που είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ε, προβλέπεται να αρχίσει σε 35 λεπτά, οπότε διακόπτουμε για 35 λεπτά. Θα αρχίσουμε όμως έγκαιρα, έτσι ακριβώς την ώρα μα. Να το ξέρετε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πολύ σύντομα.

Dear colleagues, start. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Είμαστε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, είναι το σημείο αριθμός 8, ανταλλαγή απόψεων με τον καθηγητή Νίλ Στίγεσεν, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Πρώτα απ' όλα σας καλωσορίζω εδώ κύριε καθηγητά. Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο δημιουργήθηκε μετά από την έκθεση των πέντε σοφών για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής ε, Ένωσης. Ο ρόλος του είναι πολύ σημαντικός όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, για την παρακολούθηση των δημοσιονομικών πολιτικών και για την αξιολόγηση των μελλοντικών δημοσιονομικών πλαισίων. Στις 25 Ιουλίου του 2019 δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το Γενικό Προσανατολισμό για τις δημοσιονομικές πολιτικές στην Ευρωζώνη για το 2020. Και αυτήν ακριβώς την έκθεση θα μας παρουσιάσει ο καθηγητής τώρα. Έχουμε 60 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα ακούσουμε πρώτα την εισαγωγή του καθηγητή Τίγεσεν. Υπάρχει και μια παρουσίαση PowerPoint και μετά θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Και αν ε, στο τέλος έχουμε χρόνο για κάτι Eye, θα το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλώς ορίσατε και έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι και πάλι μαζί σας, κύριε Νίντερ Μάγερ. Συγχαρητήρια σε όσους εξελέγησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάλι. Λοιπόν, τρία χρόνια υπάρχουμε τώρα, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο δηλαδή, και πάντα ήταν χαρά μας να βρισκόμαστε εδώ στην Επιτροπή σας και με τον κύριο Γκουαλτιέρη προηγουμένω, τον Πρόεδρο, και τώρα με εσάς. Σεβουλεύουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δημοσίω όμω, γιατί παίρνουμε το λόγο σε διάφορα φόρα, όπω για παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ΕΚΟΦΗΝ και σε άλλε επίσημε ομάδε πρέπει να κοιτάμε πώς πάει ο δημοσιονομικός προσανατολισμός στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Εδώ υπάρχουν κάποιες διαφάνειες οι οποίες ε, δείχνουν πρώτα απ' όλα τον ε, Ιουνίου Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό ε, Συμβούλιο έκανε μια αξιολόγηση για τους δημοσιονομικούς προσανατολισμούς στην ε, Ευρώπη και στις χώρες μέλη. Είναι κάτι που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο, συστήθηκε με την Επιτροπή τον Νοέμβριο και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Ιανουάριο. Θα εγκριθεί μάλλον από το Συμβούλιο. Ο κύκλος αυτός βέβαια λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο. Εμείς προσπαθούμε να επισημάνουμε ε, τα δύναμα σημεία του κύκλου. Υπάρχουν και κάποια αρκετά όρατα. Όταν δημιουργήθηκε το Μάστριχ, τότε είχαμε κανόνες που θα εφαρμόζονταν στις χώρες μέλη, στα εθνικά συστήματα και όχι σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Όμως τελικά αναρωτηθήκαμε μήπως θα έπρεπε όλες αυτές τις συστάσεις που κάνουμε για τις επιμέρους χώρες να τις συγκεντρώσουμε, να δούμε τι αποτέλεσμα μπορεί να δώσει ένα καλό πολιτικό μείγμα υπό μια κεντρική αρχή. Στο διάλογο αυτό πάντως για το μείγμα πολιτικής έχει βέβαια κάποιες ε, ασυμμετρίες που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν και εκείνη κυρίως συνολικά εξετάζει το θέμα της οικονομίας στην Ευρωζώνη. Είναι στο Συμβούλιο οι υπουργοί που μπορούν να εξετάσουν καλύτερα τι γίνεται σε κάθε χώρα. Θα δείτε πάντως ότι και το Συμβούλιο αντιμετωπίζει δυσκολίες. Λοιπόν, οι συστάσεις δίνονται. Εδώ έχουμε την έκθεση που αφορά το σενάριο του 2020 και βασιζόμαστε σε εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενημερώθηκαν κάπως με τις προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο. Πρόκειται για την οικονομική δραστηριότητα που φαίνεται ότι μειώθηκε από τις αρχές του 2019. Αλλά μετά από την αδυναμία αυτή υπάρχουν προοπτικές για ε, παρετέρω ανάπτυξη στο δεύτερο εξάμεινο του 2019 και καλύτερες επιδόσεις το 2020. Αναγνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι στις προπτικές οι οποίοι γίνονται όλο και πιο σημαντικοί εξαιτίας του Brexit, εξαιτίας εμπορικών εντάσεων και προβλημάτων στην μεταποίηση. Η επόμενη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα γίνει τον Νοέμβριο, οπότε το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο πρέπει να κάνει μια ανεξάρτητη εκτίμηση. Βασιζόμαστε στις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά τίποτα παραπάνω. Εδώ είναι οι εικόνες που μας βοηθούν να προβούμε στις δικές μας εκτιμήσεις. Και παρά τις ε, σκοτεινές προοπτικές, η απασχόληση βελτιώνεται, η ενεργεία μειώθηκε δηλαδή και, και θα εξακολουθεί να μειώνεται και το 2020 βάσει των προβλέψεων και μια ανάπτυξη 1,1-1,2%. Κάτι που ευθυγραμμίζεται και είναι λίγο παραπάνω από τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης, τη δυνητική ανάπτυξη δηλαδή. Εδώ βλέπετε τους δείκτες για τις διάφορες χώρες. για τις χώρες της Ευρωζώνης και γενικά τις 28 χώρες ε, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ βλέπουμε την ίδια πορεία με μείωση αλλά με κάποια ε, συμμετρία για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Στην Ευρωζώνη δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει το συνολικό από τα επιμέρους συστατικά. Εδώ έχουμε τα σύνολα. και δείχνει σε τι βαθμό ήταν προκυκλικές οι πολιτικές και σε, βαθμό, σε τι βαθμό ήταν αντικυκλικές κατά το παρελθόν. Και εδώ βλέπουμε ότι υπήρξε μια συστολή και μετά την κρίση από το 2011 μέχρι το 2013 δηλαδή. Μια έντονη περίοδος προκυκλικής πολιτικής, αντίθεση με το 2014 με 2018, όπου ο, φορολογικός, ο, συγνώμη, ο δημοσιονομικός προσανατολισμός ήταν διαφορετικός. Και για το 2019 και 2020 βλέπουμε ότι μπαίνουμε σε μια μεγαλύτερη επέκταση. Ε, δεν έχουμε πια το κενό αυτό το χάσμα παραγωγής και βλέπουμε ότι τα επίπεδα ανάπτυξης είναι θετικά. Τώρα, ο δημοσιονομικός προσανατολισμός. Πρέπει εδώ να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στους αυτόματους σταθεροποιητέ και τις ε, διαφοροποιημένε δράσεις πολιτικής που επηρεάζουν τις αποφάσεις, τι πολιτικές της χώρες μέλη. Τώρα, οι προοπτικές για το 2020. Εδώ συστήνουμε μία νέα ε, δημοσιονομική ε, προσέγγιση. Εδώ έχουμε ε, συστάσεις για ενίσχυση 0,3% του διαρθρωτικού, του βασικού ελλείμματος. Και για τις χώρες όπου έχουν μεγάλο έλλειμμα λέμε ότι μια καλή πολιτική θα ήταν να παρακολουθήσουμε από κοντά τις χώρες, να συμμορφωθούν με τις συστάσεις και χώρες που έχουν περιθώρια με πλεονέσματα να φροντίσουν αντίστοιχα την πολιτική τους, να δαπανίσουν δηλαδή. Εδώ βλέπετε τις πράσινες και τις κόκκινες ε, βούλες. Οι χώρες που είναι στις κόκκινες βούλες έχουν υψηλά ελλείμματα. Είναι πέντε που έχουν εντοπιστεί σε αυτή την ομάδα. Και είναι αυτές που έχουν περισσότερες πιθανότητες επέκτασης. Υπάρχουν τώρα άλλες χώρες οι οποίες έχουν πλεόνασμα και θα μπορούσαν να ξοδεύουν περισσότερα. Έχουν δηλαδή προπτικές, αλλά δυστυχώς μόνο πολύ μικρό ποσοστό του δημοσιονομικού του περιθωρίου χρησιμοποιούν αυτές οι χώρες όπως η Γερμανία. Θα έπρεπε να κάνουν περισσότερα. Στρεφόμαστε τώρα στους καθοδικούς κινδύνους οι οποίοι αναδύονται και πιστεύω ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτά που είπε χτες ο πρόεδρος Ντράγκη. Υπενθυμίζω ότι σε μία επιβράδυνση όπως έχουμε τώρα, γιατί έτσι εγώ θα περιέγραφα το 2019 και 2020, αυτόματοι σταθεροποιητές ε, λειτουργούν, θα λειτουργήσουν και μερικές φορές θα κάνουν τις χώρες να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες. Αλλά η κύρια φιλοσοφία του Μάστριξ στο κάτω-κάτω είναι ότι αν παρακολουθείς συνετές πολιτικές και φροντίσεις τις διευθυντικές σου πολιτικές και το έλλειμμά σου, τότε μπορείς να επιτρέψεις τους αυτόματους σταθεροποιητές να λειτουργήσουν στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ιαπωνία. Οι σταθεροποιητές αυτοί είναι περισσότερο ισχυροί. Πάντως δεν είναι κάτι που πρέπει να παραβλέπουμε. Τώρα δεν φτάνει. Υπάρχουν αρκετά αρνητικά στοιχεία σε αυτό το σενάριο, γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ευελιξία στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η προσαρμογή αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί από διάφορες χώρες στις δραστηριότητές τους. Την ευελιξία αυτή βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα την ερμηνεύσουμε, όπως έγινε το 2015 που ήμασταν επικριτικοί γιατί υπονομεύω τους κανόνες μερικές φορές. Όμως, αν χρειαστεί, πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η ευελιξία. Υπάρχει βέβαια και μια ρήτρα εξαίρεση σε περίπτωση μεγάλης οικονομικής ύφεσης. Ναι, οι κρίσεις. Πιστεύουμε ότι τα αρνητικά στοιχεία που έχουμε στις προοπτικές δεν ε, μας επιτρέπουν να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη ρήτρα εξαίρεσης. Πάντως, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο πιστεύουμε ότι η κεντρική δημοσιονομική ικανότητα χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν ε, σύγχρονες αναταράξεις και όχι μη συμμετρικές. Τι χρειαζόμαστε αυτή την κεντρική δημοσιονομική ικανότητα. Από την άλλη υπάρχουν κάποια στοιχεία ε, τα επόμενα χρόνια για τη σύγκληση που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μια πρόσφατη έκθεση, και δεν τη συζήτησα την προηγούμενη φορά, γιατί έχει να κάνει με την επόμενη έκθεσή μας, που θα σταλεί και στη δικιά σας επιτροπή, με την ετήσια έκθεσή μας, έχουμε εξετάσει τους κανόνες Και εδώ συζητάμε την ισορροπία ανάμεσα στην ελαστικότητα και την σταθεροποίηση, προκειμένου να έχουμε ε, υγιή δημοσιονομικά. Θα σταματήσω εδώ, Πρόεδρε, και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Σας ευχαριστώ. Ελπίζουμε να είμαστε τόσο οργανωμένοι όσο και εσείς. Σας περάσουμε τώρα τις ερωταπαντήσεις. Παρακαλώ μπορείτε να διατυπώσετε με σαφήνεια τις ερωτήσεις σας, για να έχουμε και αρκετό χρόνο για τις απαντήσεις και να μπορέσουμε να σεβαστούμε και το χρόνο μέσα σε πέντε λεπτά από το έλκο. ο κύριος ε, Στέφαν Πέρκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά. Κύριε Τιγκέζεν, εμείς ε, από το ΕΛΚΑ συμφωνούμε με την ανάλυση που κάνατε. Στην τελευταία διαφάνεια που δεν τη διαβάσατε, εκεί ε, κατ' ουσίαν υπάρχει ε, μια ολόκληρη δέσμη μέτρων ε, μια μέτρων που δημοσιοποιήσατε την προηγούμενη εβδομάδα. Σκεφτόσατε λοιπόν, σκεφτόσαστε να εισαγάγετε στην Ευρώπη ένα χρυσό κανόνα ε, χρυσός κανόνας πάντα είναι μία δικαιολογία για να μπορεί κανείς ε, να κάνει περισσότερα χρέη. Η συμπεριφορά των κρατών μελών, το είπατε κι εσείς, ε, είναι διαφορετική. Στη Γερμανία ισχύει το απόλυτο μηδέν, εκεί δεν γίνονται χρέη. Σε άλλες χώρες όμως η πολιτική δαπανών είναι τελείως διαφορετική. Και ε, ρωτώ, αν έχει κανείς ε, κατά νου το χρυσό κανόνα, τι είδους επενδύσεις έχετε κατά νου που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα τέτοιο χρυσό κανόνα. Και ένας ε, χρυσός κανόνας δεν θα επηρέαζε την δημοσιονομική πολιτική και πειθαρχία στην Ευρώπη. Δεν θα την υπονόμευε. Και ρωτώ, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί ή μήπως ε, δεν θα συγκέντρωνε την απαραίτητη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ε, είναι μια ερώτηση που ετέθη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο άτυπο Συμβούλιο Εκοφήν. Ο χρυσός κανόνας είναι ένας τρόπος για να προστατευτούν οι επενδύσεις. Ένα πρόβλημα με τους ε, δημοσιονομικούς κανόνες, ε, τώρα που κοιτάμε προς τα πίσω την κρίση, είναι το ότι οι κυβερνήσεις περιορίζουν κατά κύριο λόγο τις επενδύσεις ε, στην κρίση. Δηλαδή προστατεύουν άλλα αγαθά, τους δημόσιου μισθού, την κατανάλωση, αλλά αλλά ε, η περικοπή των επενδύσεων είναι και το βασικό αίτιο της βραδίας ανάπτυξης που έχουμε σήμερα στην Ευρώπη. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες ε, ρήτρες περί αλλά ε, μόνο οι χώρες που έχουν αυτό το κενό του 1,5% μπορούν να καταφύγουν σε αυτή τη ρήτρα. Αυτό έγινε πρόσφατα από την Ιταλία οι χώρε θα έπρεπε να το σκεφτούν λιγάκι περισσότερο. Όσον αφορά το χρυσό κανόνα, εδώ υπάρχουν διτά προβλήματα. Ε, τι είδου επενδύσει εμεί λέμε στην δική μα την αξιολόγηση ότι θα πρέπει να είναι στοχευμένε ε, να είναι στοχευμένες ε, σε επενδυτικά αγαθά που έχουν προτεραιότητα. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα όπου οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να συμβάλλουν. Εάν συμβάλλουν περισσότερο από ό,τι προβλέπεται, αυτό θα μπορούσε να είναι μια αποδοτική επένδυση. Στον τομέα της κλιματικής αλλαγής υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες ε, Άρα δηλαδή η στόχευση είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Ο δεύτερος στόχος είναι η συνθήκη του Μάστριχτ, το πώς αντιμετωπίζονται ε, τα χρέη και τα ελλείμματα ε, και να μην λένε αυτό που λένε οι περισσότερες κυβερνήσεις ότι οι δαπάνες είναι δική μας υπόθεση. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να πιστούν οι κυβερνήσεις και ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες αλλαγές των δημοσιονομικών κανόνων. Αλλά πολύ σωστά ε, προβληματίζεστε για την υπονόμευση των κανόνων, γιατί ε, εισάγονται νέοι περίπλοκοι κανόνες. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτεροι από ό,τι άλλοι που υπήρχαν κατά το παρελθόν. Γιώνας Φερνάντες από τους Σοσιαλδημοκράτες. Καλώς ήλθατε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τη σύσταση σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη και τη συνολική δημοσιονομική θέση. Εσείς συστήνετε ουδετερότητα. Σε ποιο βαθμό αυτή η ουδετερότητα της δημοσιονομικής πολιτικής θα έκανε την ΕΚΤ να έχει μια πιο επεκτατική νομισματική πολιτική από αυτή που τη συμβουλεύουν ή επαρκώς ε, για να προκαλέσει προβλήματα μεσονομική ε, σταθερότητα, όπως ακούσαμε χθε από τον κύριο Τράγκη. Και για να διορθώσουμε αυτά τα προβλήματα, ίσω θα μπορούσε να είναι άλλη δημοσιονομική θέση, επειδή οι προβλέψεις ε, για του χρόνου δεν είναι και τόσο θετικές, ε, όπως δεν ήταν όπως και κάποιου μήνε πριν. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά την κατανομή αυτής της ουδέτερης θέσης της δημοσιονομικής πολιτικής σε ποιο βαθμό αυτή η ουδέτερη πολιτική που υπερασπίζεστε σε καθολικό επίπεδο της Ευρωζώνης, πώς θα καταναμηθεί μεταξύ των διάφορων κρατών, έτσι ώστε κάποιοι θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν προσπάθειες ε, για να σταθεροποιήσουν, να εξηγιάνουν τους προπολογισμού τους, ε, ενώ κάποιοι άλλοι θα ε, μπορούσαν να μας πείτε τι θα μπορούσαν να κάνουν για να πετύχουν τουλάχιστον αυτή την ουδέτερη δημοσιονομική στάση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φερνάντες για τις ε, δύο ερωτήσεις. Είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση σήμερα. Είμαι αρκετά μεγάλος για να έχω συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ε, του Μάστρικτ ε, και τότε έλεγε η ΕΚΤ ότι θα πρέπει να την προστατεύσουμε κατά των κυβερνήσεων με υψηλό χρέος και υψηλές δαπάνες, έτσι ώστε να μην πιέζουν την Κεντρική Τράπεζα να διατηρήσει χαμηλά επιτεόκια για να εξυπηρετεί χώρε με υψηλό χρέο. Σήμερα έχουμε χώρε με υψηλό χρέο, αλλά έχουμε μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που το ζητά να κάνουν περισσότερο παρόλα αυτά. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η δική σα κατάσταση που αιτιολογείται από την ε, αλλαγή στην προοπτική και από το γεγονός ότι είναι ανεξάρτητο όργανο τώρα η ΕΚΤ. Βέβαια, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο είχαμε συζητήσει το 2014 καταρχήν όταν ο κύριος ε, Ντράγκη μίλησε για απαραίτητο μείγμα πολιτική και ότι οι δημοσιονομικές αρχές πρέπει να κάνουν περισσότερα για να αποφύγουν τον αποπληθωρισμό και ε, σήμερα πρέπει να κάνουν περισσότερο και πρέπει η ΕΚΤ να φτάσει το στόχο σχετικά με τον πληθωρισμό. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρου τη ΕΚΤ πόσο περισσότερο μπορεί να κάνει, πρέπει να κάνει για να είναι ενεργός η δημοσιονομική πολιτική. Όμως τα όσα μας είπαν συνάδουν με τις παρατηρήσεις της δικές μας ότι χρειάζονται κάποια δημοσιονομικά κίνητρα και εντός της Ευρωζώνης. Η ουδετερότητα δεν σημαίνει ότι πρέπει να τηρηθεί από όλου. Σε κάποιες χώρες που υπάρχει δημοσιονομικός χώρος μιλάμε και για επέκταση. Και έρχομαι τώρα στο άλλο ερώτημα. Νομίζω ότι αυτό είπε και ο κύριος Ντράγκη. Οι χώρες με πολύ ψηλό χρέος θα πρέπει και πάλι να ασκήσουν σόφρονες πολιτικές και ίσως ε, φέτος ή του χρόνου να μην μπορούν να συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πρόγραμμα. Αυτό ε, ε, το είδαμε το 2019 όταν ανέστηλε η Κομισιόν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ουσιαστικά. Αυτή ήταν πολύ ωραία ιδέα, αλλά δεν διαφοροποιούταν επαρκώς μεταξύ των χωρών. Και κάποιες χώρες με αδύναμα οικονομικά Επίσης, ε, ε, συμμετείχαν και είχαν πάρα πολύ δύσκολη περίοδο γιατί είδαν περαιτέρω αποδυνάμωση. Τώρα, η πρόκληση είναι να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση για να έχουμε ένα πολύ προσεκτικό μείγμα παροχής συμβουλών. Εδώ δεν το διευκρινίζουμε. Απλώς ε, λέμε ότι μπορεί να υπάρχει ο χώρος και είδατε το διάγραμμα στη διαφάνεια. Μας δείχνει ποιες είναι οι αποστάσεις μεταξύ των δημοσιονομικών χωρών στις μεμονωμένες χώρες. Μπορείτε να το εξετάσετε κι εσείς στις διαφάνειες. Υπάρχει λοιπόν διαφοροποιημένη συμβουλή που μπορεί να δοθεί εδώ. Δεν ε, υπάρχουν αριθμιστικά στοιχεία να αναφερθούν αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καρκάνου για το Ρινιού. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστούμε κύριε Τίτσεν, που είστε εδώ. Όπως και άλλοι, εγώ διάβασα την εκθεσή σας και την αξιολόγησή σας και με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τη σημερινή σας παρέμβαση. Η αξιολόγησή σας ήταν, όπως ε, είπατε, ότι χρειαζόμαστε εργαλεία για να έχουμε ένα συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό για να αντιμετωπίσουμε τα σοκ και θα πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από τις ε, συμβουλές που δίνονται. Θα ήθελα όμως, ε, αν είναι δυνατόν, να μπούμε και στο θέμα των μεταρρυθμίσεων και των ε, θεσμικών οργάνων. Βασικά, εν μέρη, θα βασιστώ σε αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος. Καταρχήν, χωρίς κοινό δημοσιονομικό εργαλείο, όπως ένας ε, αντικυκλικός προπολογισμός της Ευρωζώνης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Πώς ε, η Ευρώπη, πώς ε, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες που πρέπει να έχουν μία πιο επεκτατικό δημοσιονομικό προσανατολισμό. Το θα πρέπει να υιοθετηθεί από τη Γερμανία και την Ολλανδία, παραδείγματος χάρη είπατε. Φαίνεται ε, ότι έχουμε ένα ε, παλιό πρόβλημα ότι ασύμετρα εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες ε, και από τις χώρες που είναι σε Τώρα έχουμε νέα πρόταση από, το νέο, τη νέα πρόεδρο της Κομισιόν προκειμένου να έχουμε αυτό τον συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό και να υπάρχει ένας μηχανισμός αντασφάλισης πιστεύετε ότι αυτός ο μηχανισμός είναι ένας τρόπος να εκφραστεί αυτό, είναι επαρκής, είναι ένα καλός τρόπος να προχωρήσουμε και πιστεύετε ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι στόχος. Μιλάτε στην εκθεσή σας για τις επενδύσεις. Ποιο θα είναι, ε, το, ποιο θα είναι το ιδανικό ε, συνολικό εργαλείο που προτείνετε εσείς. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με τη δεύτερη ερώτησή σας ε, για τον μηχανισμό που αφορά την ανεργία. Αυτός ο μηχανισμός έχει συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό και εμείς έχουμε δώσει συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς να δημιουργήσουν ε, δημόσιους ε, μηχανισμούς χρηματοδότησης από το 1973, αν ε, το πιστεύετε. Είχαμε διάφορες ομάδες συζήτησης και η κύρια ιδέα ήταν ένα ταμείο ασφάλισης για την ανεργία. Νομίζω ότι η Κομισιόν ε, έχει σχεδιάσει κάτι τέτοιο, ε, καθορίζοντας ποιο είναι το επίπεδο. Ε, πρέπει να έχει σε ψηλό επίπεδο απασχόλησης και ένα στόχο πέρα από αυτό. Ίσως να έχει δοθεί υπερβολική έμφαση μακροπρόθεσμα στο θέμα της αποπληρωμής αυτού του μηχανισμού, όμως υπάρχει ένα πολιτικό τίμημα που πρέπει να πληρώσει κανείς αυτό φαινόταν ως ένα κεντρικό στοιχείο ε, στα πλαίσια της δημοσιονομικής ικανότητας να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός και νομίζω ότι θα είχε κάποια πλεονεκτήματα. Εμείς στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό είδαμε ότι δινόταν υπερβολική έμφαση μόνο στην ιδέα των ασύμετρων σοκ που υπάρχουν από την απαρχή της Ευρωζώνης. Ε, υπάρχει ένας μηχανισμός αναδιακατανομής, ανακατανομής, όμως μερικές φορές έχουμε κοινά σοκ και τότε θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε μία ικανότητα, ένα μηχανισμό. Έγινε αυτό το 2008-2009 και βλέπουμε ότι η Γερμανία και η Ιταλία για μια φορά είναι δύο χώρε που φαίνεται να εκτίθενται περισσότερο σε αρνητικό σοκ. Δεν έχουμε ένα σύμμετρο σοκ σε μια χώρα μόνο, αλλά αφορά ολοκλήρη την Ευρωζώνη, αν μιλάμε για τέτοιο σοκ. Έτσι λοιπόν νομίζω ένας ε, μηχανισμός ε, τέτοιος είναι μόνο ένα πράγμα που έχουμε συζητήσει και αν το έχει στο πρόγραμμά τη ε, η πρόεδρο τη Κομισιόν θα ξανασυζητηθεί. Όμω θα πρέπει να συμπληρωθεί και από άλλα στοιχεία σε ό,τι αφορά μια κεντρική δημοσιονομική ικανότητα. Τώρα, πώς, είπατε πώς θα πείσουμε τις χώρες ε, που είναι κάπως διστακτικές. Οι χώρες που βρίσκονται σε δυσκολία ε, θα πρέπει να δουν ε, πώς μπορούν να βγουν από την ύφεση. Όμως πώς θα το κάνουν οι χώρες που έχουν πλεόνασμα δεν μπορείς ακριβώς να τους το υποδείξεις οι δείκτες ε, μας δείχνουν ότι έχουν υψηλά ποσοστά αποσχόληση. Τώρα η Γερμανία έχει ένα αρνητικό κενό output, ε, όμως φαίνεται ότι αρχίζει να σκέφτεται πολύ προσεκτικά επί του θέματος και θα υπάρχουν εξέλιξεις στη Γερμανία, όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι με τους σημερινούς κανόνες είναι θέμα πειθούς περισσότερο, παρά εφαρμογή κανόνων. Όμως, ε, υποκείμενη κατάσταση έχει ήδη οδηγήσει σε κάποια αναθεώρηση του σκεπτικού και στις κατοχώρες και στη Γερμανία και πιθανότατα και, άλλες χώρες, και σε άλλες χώρες που έχουν τέτοιο δημοσιονομικό χώρο. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες από τα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ. Όταν συναντηθήκαμε, ο κύριος ε, καθηγητής μου είπε ότι είχαμε συναντηθεί πριν από 20 χρόνια στην Κεντρική Τράπεζα στην ε, Πράγα. Ε, και βλέπω τώρα ότι πάει πίσω στο 73-74 και θυμάται πράγματα πραγματικά απίστευτο. Ο κύριος Ούρτανσον από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά που ήρθατε σήμερα. Όσον αφορά την έκθεση, για το ενδεχόμενο αναθεώρηση των κανόνων. Ένα από τα πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αν αναλύσει κανείς ε, την συνεχή ε, προκυκλικότητα των κανόνων, στην έκθεση βλέπουμε ότι από το 90 μέχρι το 2018 υπήρξε μόνο μία βασική αντικυκλική επέκταση ε, το 9. Τότε ήταν το πρόγραμμα της οικονομικής ανάπτυξης και τότε προκυκλική επέκταση με, την, με το ευρώ το 2000 και μία άλλη προκυκλική εξέλιξη από το 11 μέχρι το 2013. Άρα δηλαδή είναι απόλυτα σαφές ότι βρισκόμαστε μέσα από το πλαίσιο των προκυκλικών κανόνων και θέλουμε να μας εξηγήσετε πώς κατά την άποψή σας πρέπει να εξηγήσουμε αυτή την προκυκλική ε, κατεύθυνση και εξέλιξη και τι σημασία έχουν οι κανόνες. Η δεύτερη ερώτηση είναι περισσότερη, ε, έχει σχέση με τη μέθοδο. Ε, στις συστάσεις πολιτικής που κάνουμε υπάρχει μία έννοια που είναι πολύ σημαντική και είναι το, οι ενδεχόμενες εξελίξεις, το αποτέλεσμα, η παραγωγή. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας ερωτήσω. Αυτό δεν πιστεύετε και εσείς ότι θα πρέπει να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στις προβλέψεις που κάνουμε σχετικά με την προτινόμενη πολιτική. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δύο ερωτήσεις. Έχετε ε, απόλυτα δίκιο σε αυτό που είπατε σχετικά με την προκυκλικότητα. Αυτή είναι μια ιστορία επιτυχίας ε, η επέκταση μετά το 9, το 9-10, τότε σωστά πράξαμε. Βέβαια, τρία χρόνια προκυκλικότητες ανησυχούν. Και πάλι εδώ υπάρχει μια ασυμμετρία που είναι ε, πολύ δύσκολο να αποφευθεί, να πιστούν δηλαδή οι χώρες σε καλές εποχές, να προβαίνουν σε σταθεροποίηση και να έχουν αντικυκλικές πολιτικές όταν ακριβώς τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Αυτά αναφέρονται ε, και στην έκθεσή μας που μόλις τώρα ολοκληρώσαμε το 2018. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Πώς μπορεί κανείς να προετοιμαστεί ε, εγώ θα έλεγα τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Η επιτυχημένη ιστορία δεν διαχύθηκε αρκετά. Ε, το 1113, ένα μέρος της προκυκλικότητας ήταν όχι μόνο δημοσιονομικό, αλλά ήταν σαφώς η υποτίμηση των επιπτώσεων της ε, παράλληλης ε, συρρήκνωσης. Κανείς δεν ήξερε τι θα γίνει μετά τη βαθιά κρίση. Άρα δηλαδή όχι άμεση σχέση με τους κανόνες, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο ε, προβλέφθηκε το όλο αυτό σύστημα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πήγαν στραβά και εγώ πιστεύω ότι η νομισματική πολιτική μέχρι το 2011 δεν συνέβαλε με τον ίδιο τρόπο όπως σε άλλες περιοχές του κόσμου για να αμβληθούν οι επιπτώσεις ε, του αρνητικού σοκ. Στην πρόταση για μεταρρύθμιση εισάγουμε κατά κάποιον τρόπο αναδιατύπωση των κανόνων της εξυπηρέτησης του χρέους, ε, να υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο περιθώριο για αντικυκλικές ε, πολιτικές για μία ετών. Ε, όσον αφορά την έκθεσή μου και το προβλέψετε ήδη, είναι μια μακροσκελής έκθεση που ε, δεν μπορώ να παρουσιάσω στην Επιτροπή. Ας παραμείνουμε προς τα ε, προς το παρόν εκεί. Όσον αφορά τώρα τις προβλέψεις, θέλω να πω ότι οι κανόνες, επειδή βασίζονται στην έννοια της ε, παρατήρησης που είναι καθοριστική και για το έλλειμμα, προσφέρει μια απίστευτη ισχύ ε, των κανόνων που αυτό όμως μακροπρόθεσμα επιζήμιο. Ο υπερτονισμός δεν είναι κάτι το απαραίτητα θετικό. Εμείς λοιπόν προτείνουμε στις μεταρρυθμίσεις να καταργηθεί το μη απορροφούμενο και να περάσουμε μόνο σε ό,τι μπορεί να απορροφηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αυτό προφανώς είναι πάρα πολύ ριζικό για πάρα πολλές χώρες. Ως οικονομολόγος θέλω να πω ότι ε, το ενδεχόμενο του αποτελέσματος είναι καλό ως ε, αναλυτικό στοιχείο. Είναι δύσκολο βέβαια να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα ε, γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν απορροφήσει τους κανόνες και άλλες που λένε ότι δεν τους λαμβάνουμε παρκώς υπόψη μας. Δεν υπάρχει κανείς από την πολιτική ομάδα ID. Το ECR δεν ήθελε να λάβει το λόγο. Άρα πάω τώρα στην Κουη, η κυρία Ομπρή. Δεν ξέρω αν κάθομαι στη σωστή θέση, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ κάθομαι τώρα. Γαλλικά θα μιλήσω. Πρώτα απ' όλα καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ για την έκθεσή σας. Δεν είχα εγώ την τύχη πριν από 20 χρόνια να σας συναντήσω, αλλά έχω την ευκαιρία και θα έχω και στο μέλλον την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψη μαζί σας για την έκθεση αυτή. Υπάρχουν πολλά συμπεράσματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τρία ως επιτοπλίστων. Πρώτον, διαβάζοντας την έκθεσή σας βλέπω ότι ενώ τα κριτήρια σύγκλησης αναφέρονται συχνά από τους επικεφαλεί κατών και κυβερνήσεων για να δικαιολογήσουν τη λιτότητα. Τα ξέρουμε όλοι αυτά στις χώρες μας. Η έκθεσή σας μιλάει για την περιορισμένη αποτελεσματικότητα, αν μη τι άλλο, αυτών των κανόνων λιτότητα και της δημοσιονομικής πειθαρχία γενικότερα ότι δεν οδηγούν στα αποτελέσματα που θα θέλαμε, ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες χώρες που δεν τηρούν τους κανόνες από ότι το αντίθετο και ανάμεσα στην οικονομική σύγκληση και το ευρωπαϊκό εξάμενο ε, δεν υπάρχει απαραίτητα άμεση ε, σύνδεση και πολύ έντονη. Οπότε αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον στην έκθεσή σας και θα ήθελα να τονίσω είναι τα αρνητικά που αναφέρετε και εσείς από το Ευρωπαϊκό ε, Εξάμεινο. Οι επενδύσεις κρατικές για την εκπαίδευση, τις μεταφορές, ε, ανάπτυξη κτλ. που αναγκάζουν τις χώρες να περικόπτουν στις δημόσιες δαπάνες για να τηρούν το 3%. Κάτι το οποίο οδηγεί και σε εντάσεις μεταξύ χωρών μελών. Ρωτώ λοιπόν, δεδομένων όλων αυτών, πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που έχει περιορισμένα αποτελέσματα και παρενέργειες πιστεύετε ότι πρέπει να εξακολουθεί να ισχύει. Επίσης βλέπουμε στις ε, συστάσεις σας αν αλλάξουμε τους κανόνες του ελλείμματος από κάτι άλλο, μία οροφή. Μήπως αυξήθηκε το έλλειμμα επειδή τελικά οι χώρες αναγκάστηκαν να σώσουν τις τραπεζές τους και μεταφέρθηκε το ιδιωτικό χρέος στο δημόσιο χρέος. Και αν θέλουμε να προστατεύσουμε τις δημόσιες δαπάνες όπως λέτε, τότε γιατί από την οροφή κρατικών δαπανών να αφαιρέσουμε προγράμματα και σχέδια που είναι προς όφελος της Ευρώπης. Και έπειτα εσείς λέτε γιατί όχι η οικολογική μετάβαση. Μήπω και αυτές οι δαπάνες που πηγαίνουν για την οικολογική μετάβαση θα έπρεπε να αφαιρούνται από τα κριτήρια που ορίζουν το χρέο και το έλλειμμα. Απάντηση. Η αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών κανόνων είναι μια δύσκολη έννοια γιατί οι στόχοι είναι αντιφατικοί μερικές φορές. Έχουμε πει ότι υπάρχουν τρία κριτήρια για την αποτελεσματικότητα αυτή. Το ένα είναι η βιωσιμότητα, υπάρχει βιωσιμότητα. Το δεύτερο ήταν επιτρέπουν αντικυκλικές ε, πολιτικές και αποφεύγουν προκυκλικές. Και το τρίτον συνεισφέρουν στην ποιότητα των ε, δημοσίων δαπανών. Αυτά τα τρία στοιχεία οδηγούν σε διαφορετικές απαντήσεις όταν προσπαθεί κανείς να κρίνει την αποτελεσματικότητα. Ένα στοιχείο ήταν ότι στην νομοθεσία του 2012 και 2012 το πακέτο των 6 και το πακέτο των 2 οδηγιών, η βιωσιμότητα δεν ήταν απαραίτητα κριτήριο. Είχαμε τις αντιδράσεις των αγορών, τους δημοσιονομικούς κινδύνους, τα προβλήματα με τις τράπεζες κλπ. Και σε αυτά έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα. Έγιναν κάποιες εκτιμήσεις που τις ανέφερα και πριν για μεγαλύτερη ανάγκη για προκυκλικές περιόδους. Πάντως, υπήρξαν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που σχετίζονται με την βιωσιμότητα. Τώρα είμαστε στο 1% ενώ είμαστε 6% πριν από 10 χρόνια. Άρα οι κανόνες συνεισφέρουν. Τώρα ότι είναι περιορισμένη η αποτελεσματικότητά τους, θα σας πω το ίδιο για την προκυκλικότητα. Οι κανόνες δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικοί. Ίσως θα έπρεπε να δούμε την νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να δούμε συνολικά τους κανόνες και όχι μόνο να μιλάμε για απλοποίηση. Και εκείνοι αναγνωρίζουν ότι οι κανόνες έχουν γίνει πολύ περίπλοκοι και κατά μία έννοια και αναποτελεσματικοί. Τα δύο λοιπόν ισχύουν, το τρίτο όχι. Γι' αυτό και προτείνουμε το χρυσό κανόνα για να προστατεύουμε τις επενδύσεις εκείνες που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Και πάμε έτσι και σε άλλες προτάσεις που έγιναν από το Ζακ Ντελόρ, για παράδειγμα, τότε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, υιοθετούμε μία παλιά ιδέα δεν μιλάμε μόνο για απλοποίηση. Αλλά δεν πρέπει να έχετε και την ε, ψευδέστηση ότι μπορεί οι δημοσιονομικοί κανόνες να εξυπηρετούν ε, κάθε σκοπό. Χρειάζονται διάφορα εργαλεία ανάλογα με τους στόχους και σίγουρα τα δημοσιονομικά εργαλεία δεν μπορούν να πετύχουν ε, όλους τους στόχους, όποιο και αν είναι το αντικείμενο. Περνάμε στο Κατσιδιάη, ο κύριος Μάρκες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Παρακολούθησα την παρουσίασή σας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βασικά μας είπατε ότι έχουμε κλείσει το κενό ε, των οικονομικών επιδόσεων αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Όμως ε, δεν έχουμε αύξηση του πληθωρισμού, σαφέστατα. Έτσι λοιπόν, ε, από ό,τι φαίνεται, δεν υπερτροφούνται την ευρωπαϊκή οικονομία. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Είμαστε παγιδευμένοι σε έναν φαυλοκύκλο χαμηλή ανάπτυξη για πολύ καιρό και το ίδιο μάλλον θα ισχύσει και στο μέλλον. Αυτό είναι ένα κίνδυνο για την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν παράγουμε αποτελέσματα, δηλαδή δεν δημιουργούμε συνθήκες για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών και να αυξήσουμε τα εισοδήματα των πολιτών ε, με έναν ε, σημαντικό τρόπο για τα επόμενα χρόνια. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι δυνητικές ε, οικονομικές επιδόσεις ή το χάσμα όπως αναφέρετε, αυτά τα μέτρα ουσιαστικά περιόριζαν την ε, ικανότητά μας να εφαρμόσουμε πολιτικές που να δημιουργούν περισσότερη ανάπτυξη για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτή η ιδέα που μας παρουσιάσατε σήμερα, ότι πιθανότατα τώρα θα πρέπει να είμαστε σε, μια πιο, ε, σε έναν πιο σόφρονα δημοσιονομικό προσανατολισμό και τις χώρες που έχουν σημαντικό πλεόνασμα. Δεν θα έπρεπε να κάνουν περισσότερα. Και θα ρωτήσω πώς το Δημοσιονομικό Συμβούλιο βλέπει τις ε, πρόσφατες ανακοινώσεις ε, της γερμανικής κοινωνικής κυβέρνησης για το δημοσιονομικό προσανατολισμό για το επόμενο χρόνο, κυρίως αυτό που αναφέρατε στην παρουσίασή σας. Και τέλος, η τελευταία σας μόλις αναφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι υπερβολικά προγεκλικό. Θα πρέπει να το αλλάξουμε λοιπόν και αναφέρατε κάποιες προτάσεις. Είπατε ότι θέλουμε σημαντική βελτίωση και όχι μικρές απλουστεύσεις. Ποια θα ήταν η πρώτη σας προτεραιότητα, θα το αλλάζετε για έναν κανόνα σχετικά με τις δαπάνες ή πώς θα το αλλάζετε σημαντικά έτσι ώστε να εγκαταλείψουμε, να εγκαταλείψουμε με συγχωρείτε αυτούς τους προκυκλικούς κανόνες. Έχετε δίκιο ότι η ευρωπαϊκή οικονομία υπερθερμαίνεται, όπως αναφέρα και πριν. Δεν δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα του καινού των οικονομικών επιδόσεων δεν είναι πλέον ένας καλός ε, δείκτης ε, για τις πληθωριστικές τάσεις και η ΕΚΤ νομίζω έχει διδακτεί Όμως, είναι γεγονός ότι δεν έχουμε αυτές τις στιγμές δημοσιονομικές ε, πολιτικές που να λειτουργούν ως προς το να τονώσουν τη ζήτηση και επομένως θα πρέπει να δούμε τις δυνητικές οικονομικές επιδόσεις, δηλαδή πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τις οικονομικές επιδόσεις στο μέλλον και να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε ε, αύξηση έχουμε στις δαπάνες ε, θα γίνεται σε τομείς που θα εξηγαίνουν τις οικονομίες μας. Θα πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τις επενδύσεις. Δεν έχει λειτουργήσει αυτό πολύ καλά στο παρελθόν. Και σίγουρα θα πρέπει να έχουμε λιγότερες προκυκλικές πολιτικές. Είπα στην παρουσίασή μου ότι ελπίζω ότι η διαφοροποίηση των συμβουλών να μην ε, αφορά μόνο τις δαπάνες, να λαμβάνει υπόψη και το θέμα της ζήτησης, αλλά να υπάρχει και μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τα έθνη. Το πρόβλημα είναι πώς μπορείς να πείσεις κάποιους δεν ε, είμαι σίγουρος ε, για το ποια συζήτηση γίνεται στη Γερμανία και στις κατοχώρες. Θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο προπολογισμός τους για το 2020. Θα είναι έτοιμος σε τρεις εβδομάδες περίπου. Φαίνεται ότι χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερο δημοσιονομικό χώρο. Αυτό ήταν προφανές την άνοιξη. Εγώ περιμένω ότι θα υπάρξει κάποια αναθεώρηση αυτών των ιδεών. Γιατί ε, ουσιαστικά υπάρχει και μία πίεση για μακροπρόθεσμες προσαρμογές. Αυτό βλέπουμε κυρίως στη Γερμανία. Εδώ προσπαθούμε να βοηθήσουμε πώς διατυπωθούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες και να οθήσουμε προς ε, το να έχουμε αντιστάθμιση των ε, δαπανών και καλύτερη κατανομή μεταξύ των χωρών. Δύο άτομα έχουν ζητήσει το λόγο για κλούνας, από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι τα σχόλιά σας είναι νομίζω τα πιο εξειδικευμένα σχόλια που έχω ακούσει στην Επιτροπή εδώ. Βέβαια, εγώ μόλις ξεκινώ τη θητεία μου. Με ενδιαφέρει το πώς ελεπιδρούν τα καινοτόμα νομισματικά εργαλεία και η πιθανή επέκτασή τους προς το να φτάσουμε σε θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες. Αυτό ε, ουσιαστικά μπαίνει έμεσα και στον πολιτικό χώρο και αυτά τα εργαλεία εντάσσονται ε, στο να υπολογίσουμε ονομαστικές ισορροπίες. Ε, δηλαδή, Βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή κατάσταση, αυτό θέλω να ρωτήσω. Και θα μπορούσε αυτό να πλήξει την ε, μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ε, ε, ευρωπαϊκής δημοσιονομικής και οικονομικής κατάστασης. Δηλαδή, βρισκόμαστε τώρα σε ένα πειραματικό στάδιο. κάποιος είπε ότι κινούμαστε στο σκοτάδι από τη σκοπιά της νομισματικής πολιτικής όμως και από τη σκοπιά της δημοσιονομικής θα μπορούσαμε να πούμε. Εσείς βάσει της εμπειρίας σας θα μπορούσατε να μας πείτε. Νομίζω ότι θα μπορούσα να σας δώσω ολοκληρή διάλεξη και δεν έχουμε χρόνο τώρα, αλλά φυσικά έχετε δίκιο. Είναι έκτακτες οι συνθήκες που ελεπιδρούν μεταξύ της ε, Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική και δεν το έχουμε δει στο παρελθόν. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ευρωζώνη, το βλέπουμε και αλλού, στην Ιαπωνία, στι Ηνωμένε Πολιτείε σε έναν βαθμό και όντως ε, χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμό και σβάθο συζήτησης μεταξύ αυτών των δύο πολιτικών. Γιατί αν θέλαμε να μπούμε σε ποσοτική χαλάρωση για τους ανθρώπους όπως ε, το αποκαλέσατε, δηλαδή να απευθύνεται σε μονομένους αποδέκτε. Έχει γίνει αυτό μερικέ φορέ από τι ε, φορολογικέ αρχέ τη ΗΠΑ, Πολιτείες, χάρη. το σχάρι, όμως εδώ το παιχνίδι είναι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Δεν ε, θέλουμε να επαναλάβουμε αυτό που έγινε το 2009 και υπάρχει ένα όριο στο πόσο μακριά θέλει να πάει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αυτά τα εργαλεία. Δεν έχουμε μπει σε αυτό το στάδιο ακόμη. Όμως φυσικά έχουμε αρκετούς οικονομολόγου που γράφουν ε, τις προτάσει αυτές και ουσιαστικά επισέργονται στο πολιτικό θεματολόγιο. Νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε προσεκτικά, αλλά βέβαια ίσως όχι σε αυτό το στάδιο. Και τελευταία ερώτηση, ε, τελευταίος αλλά προφανώς όχι έσχατος, ο κύριος Μπέλκα. Σύντομη και τεχνική θα είναι η ερώτησή μου. Να φέρατε τους αυτόματους σταθεροποιητές ε, ως ένα είδος άμυνας έναντι των εξωτερικών σοκ. Διερωτώ με, έχετε κάποια δυνατότητα να ποσοτικοποιήσετε ε, την αποτελεσματικότητα των αυτόματων σταθεροποιητών στην Ευρώπη. Δηλαδή, αυτοί οι δημοσιονομικοί σταθεροποιητές πώς μπορούν να επηρεάσουν το θέμα της ζήτησης. Δεύτερον, έχετε προσπαθήσει να ποσοτικοποιήσετε τις δημοσιονομικές ε, συνέπειες από μια ιδιαίτερα χαλαρή και βολική οικονομική πολιτική στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπέλκα, κύριε Δικητά. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Όσον αφορά τους αυτόματους σταθεροποιητές, δεν το έχουμε μετρήσει. Ε, κάποιοι ίσως το έχουν μετρήσει στην Κομισιόν, δεν έχω πρόχειρα τα στοιχεία. Στον δημόσιο τομέα, τα έλεγα με 45-50% ε, του ΑΕΠ και η ευαισθησία των δημόσιων οικονομικών στους κύκλους είναι σαφής. Ε, τα πρώτα χρόνια μετά την εισαγωγή τους ε, προσπαθήσαμε να ποσοτικοποιήσουμε τους σταθεροποιητές. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι επιτρέπουν ε, το να υπάρχουν και διαφορές ε, στο μέγεθος ε, του σταθεροποιητή. Όσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος να διολυστήσει μια χώρα σε λίμματα, τόσο πιο προσεκτική πρέπει να είναι. Υπάρχουν κάποια εργαλεία. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η σύνθεση της ζήτησης, πώς την ερμηνεύει κανείς. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις χώρες, αλλά σε γενικές γραμμές πράγματι υπάρχουν ε, επιπτώσεις, σημαντικές επιπτώσεις από τους ε, αυτόμας ανθρωπιτές, γιατί τα μισά στοιχεία περνάνε από τα δημόσια οικονομικά. Δεν ε, έχουμε κάνει κάποιες μετρήσεις για το πώς λειτουργούν οι χαλαρές πολιτικές, οι κερδοσκοπικές ε, προβλέψεις. Εγώ δεν τις αποκλείω, δεν είμαι από εκείνους που τις αποκλείουν πλήρως, αλλά η εμπειρία μας με την νομισματική πολιτική ε, το να υπάρχει πληθωρισμός του 2% αυτό μας υπενθυμίζει πολύ καλά ότι δεν είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι ε, και ακόμα και τα νομισματικά σύνολα δεν επηρεάζουν τις τιμές. Σίγουρα όχι, τα επιτόκια. Στη νομισματική πολιτική, στη δημοσιονομική πολιτική έχουμε και άλλο ένα πρόβλημα, ότι δεν έχουμε απορροφήσιμους στόχους. Η ΕΚΤ, δεν ξέρω έχει, την τελευταία ερώτηση δεν την κατάλαβα. Α, μπορείτε να την ξανακάνετε, σχετικά με το φόρο του άνθρακα, επί, τον, επί του άνθρακα. Αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο, είναι ένα ε, το οποίο ε, θα μπορούσε να βοηθήσει να συγκεντρωθούν πόροι που και αυτό ε, νομίζω ότι ξεπερνάει το ότι έχουμε εξετάσει. Πάντως, κατά τα επόμενα έτη θα κατατεθούν ε, σοβαρές προτάσεις για το φόρο επί του άνθρακα ε, που ίσως είναι και ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν ε, πολλά από τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Πάντως δεν έχω κάνει υπολογισμού. Uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για μένα η συζήτηση αυτή ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες ακροάσεις που είχαμε και πολύ χαίρομαι να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή μαζί σας κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Για σήμερα η επόμενη συνεδρίασή είμαστε, είμαστε, είναι 22 Οκτωβρίου στις 9 πρωί και απόγευμα. 2 και 3 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά και σας και τους συνεργάτες σας και ευχαριστούμε που ήρθατε να μοιραστείτε μαζί μας τις ε, απόψει σας. Προσβλέπουμε σε μια νέα συνάντηση.